Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε μαζί μας τον Επίτροπο, τον κύριο Ντεχίχτ, και έπρεπε να προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων. Και αυτό αφορά το μέλλον της εμπορικής πολιτικής η στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μας εξηγήσει πώς μπορεί η εμπορική πολιτική να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για το 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα έχει ξεκινήσει μια δημοσία διαβούλευση όσον αφορά την εκστρατεία επικοινωνία που θα γίνει γι' αυτό και θα δημορφωθεί μια πολιτική η οποία θα είναι κλειδί για την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε βιώσιμη και αηφόρο ανάπτυξη και έτσι να μπορούμε να έχουμε μια συμβολή σημαντική στην ανάκαμψη του διεθνούς εμπορίου. Οπότε και εμείς θα παρακολουθήσουμε αυτήν την ε, διαβούλευση επικοινωνώντας τώρα ως προς αυτό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να η ευκαιρία μας δίνεται σήμερα να ακούσουμε απευθείας τα μαντάτα από τον Επίτροπο κ. Ντεχίχτ για να μας πει τα θέματα του, τους στόχους του, ενώ ψηφιακής του 2020 που θα αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε και πάλι κύριε Επίτροπε που ήρθατε εδώ. Έτσι θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε απευθεία. Ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι στιγμές στιγμές πρόκλησης που έχουμε τώρα χαμηλή ανάπτυξη, αυξημένη ανεργία και άνοιγμα στο χρέος των κρατών μελών, στο έλλειμμά τους και στα δημόσια οικονομικά. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μια πολιτική η οποία δεν μπορεί πια να στηρίζεται στη βοήθεια του δημοσίου προς τις οικονομίες. Επομένως αυτή είναι η πρόκληση. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα πιο σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Θα πρέπει να γίνει η ατομομηχανή της ανάπτυξης της οικονομικής, θα πρέπει να γίνει το κίνητρο, κινητήρας για μια τέτοια ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα στην οικονομία. Εγώ είμαι πεπισμένο ότι θα πρέπει να έχουμε μια ανοιχτή οικονομία. Όμω να μην είμαστε και αφελεί, διότι η Ευρώπη δεν είναι δυνατόν να μείνει άοπλη όσον αφορά το διεθνέ εμπόριο. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε όσον αφορά κάποιε απόπειρε από εταίρου να έχουν προστατευτισμό ή ε, να περιφορήσουμε έναντι κάθε πείρασμο προ αυτή την κατεύθυνση και αυτό ο κύριο Μπαρόσο το έχει αναλάβει ε, εν ώψη τη συνάντηση κορυφή του G20. Επομένως θα πρέπει να κάνουμε μια τέτοια προσέγγιση για να εξασφαλίσουμε ότι το εμπόριο θα βοηθήσει για να υπάρχει καινοτομία ε, και αυτό να είναι στην καρδιά της πολιτικής μας συνόψης του 2020 για να πετύχουμε ανάπτυξη και απασχόληση. Όμως, όμως, πάνω απ' όλα θα πρέπει να έχουμε μια αηφόρο, μια ευφυή ανάπτυξη. Χωρίς να έχουμε μια τέτοια ανάπτυξη με γρηγόρα του ρυθμούς, τότε το, το, το, το κράτος ε, ευημερίας, το κράτος προνοίας είναι πάρα πολύ ευάλωτο. Να δούμε τι κάνουν οι εταίροι μας σε όλο τον κόσμο, να δούμε πώς μπορούμε να διαδώσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες. Τον περσμένο μήνα και συζητήσαμε ποιε θα είναι οι εξελίξει τον επόμενο μισή χρόνο. Αλλά σήμερα είμαι εδώ για να ακούσω τι δικέ σα απόψει, να μου πείτε εσεί πώ θέλετε να χαράξουμε την στατική μας για το άμεσο μέλλον. Ήδη έχουμε ξεκινήσει μια ευρεία διαβούλευση για το σκοπό αυτό και εγώ περιμένω πώς και πώς να πείτε την απόφαση, την, τις απόψεις σας γιατί τώρα έχετε ευξημένες αρμοδιότητες δυνάμεις της συνήθειας της Λισαβόνας όσον αφορά το εμπόριο. Και επομένω ε, θα προχωρήσει σε θέσπιση κάποια στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, κάτι το οποίο ξεκίνησε από το 2006. Οπότε τώρα θα ξεκινήσουμε τι ε, διαπραγματεύσει ελευθερών εμπορίου για να έχουμε ε, με Κορέα, Ασία, το ΑΣΕΑΝ, όλε τι αναδυόμενε εκεί αγορέ, γιατί όλα τα προγνωστικά λένε ότι αυτέ οι οικονομίε θα γίνουν ακόμα πιο ε, σημαντικές στο άμεσο μέλλον, οπότε και εμείς το δικό μας βάρος εκεί θα το ρίξουμε. Πάντως όπως έχουν τα πράγματα θεωρούμε ότι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα θα πρέπει να διερευνήσουμε περισσότερες ε, εναλλακτικέ και να προσπαθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο στο τμήμα του εμπορίου. Και δεν εννοώ να, να, να, να επεκταθούμε περισσότερο γεωγραφικά. Ε, για το Ρίο είπαμε ότι θα ξεκινήσουμε να με τις χώρες Μερκοσούρ. Όμως αυτό που εννοώ περισσότερο είναι να προχωρήσουμε σε περισσότερη ποιότητα, σε περισσότερο βάθος όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις με τους εταίρους μας. Επίσης, θέλω να σας πω τρία παραδείγματα. Τι θα πρέπει να διερευνήσουμε. Πρώτα-πρώτα, ε, έχουμε την πρώτη συνέπεια της ε, παγκοσμιοποίησης που είναι αυτά τα, τα τεχνητά σύνορα μεταξύ εσωτερικών πολιτικών και του διεθνούς εξωτερικού εμπορίου πρέπει να βρούμε ένα καινούριο πλαίσιο, να δούμε τι γίνεται και με τις άλλες οικονομίες που έχουν ελαχιστοποιήσει το κόστος για υπηρεσίες και ε, ε, προϊόντα εξαγωγές ε, διδάσκουν τους άλλους, καμιά φορά εμείς διδασκόμαστε από τους άλλους. Όμως, το έχουμε κάποια πρότυπα διεθνή τα οποία θα αναπτυχθούν, αυτό είναι το πιο σωστό από όλα. Δεύτερον, η στρατηγική ενόψη του 2020 της Ευρώπης ε, δίνει έμφαση σε κάποια ευφυή και βιώσιμη ανάπτυξη. Θέλουμε καινοτομία, θέλουμε πράσινες τεχνολογίες. Νομίζω ότι η εμπορική πολιτική μπορεί να βοηθήσει γιατί διευκολύνει το εμπόριο σχετικά. Επίσης, ε, μπορούμε να δούμε τι γίνεται με τις ε, υπηρεσίες της τεχνολογίας. Τα πράσινα αγαθά, όλα αυτά μπορεί να βοηθήσουν στο να διαδοθούν αυτές οι πράσινες τεχνολογίες και έτσι να αρχίσει ενάρετος κύκλος με περισσότερη καινοτομία και λιγότερες δαπάνες. Επίσης, έχουμε άλλες δράσεις επί τη βάση κάποιων γενικών αρχών, αυτών που ε, περιέχει η συνθήκη και που αντικατοπτρίζουν κάποιες ε, βασικές αξίες της ευρωπαϊκής οικοδόμησης, κράτος δικαίου, ε, αηφόρο ανάπτυξη, συνεργασία με τις χώρες, σεβασμό των, των φυσικών πόρων και των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Η εμπορική πολιτική είναι κλειδί για να προαχθούν, να διωθούν όλε αυτέ οι αξίε, οι αρχέ. Έχουμε πάρα πολλέ προσδοκίε από την εμπορική πολιτική. Γιατί σε πάρα πολλού τομεί έχουμε αναπτύξει τέτοια εξωτερική δράση. Και η κοινή εμπορική πολιτική είναι η αιχμή του δώρατο και θα πρέπει επομένω να ανταποκριθούμε σε αυτέ τι προσδοκίε. Ταυτόχρονα δε θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι δυνατόν όλα να τα λύσει η εμπορική πολιτική. Επομένως, το κρίσιμο ερώτημα είναι εσείς. Πώς θεωρείτε ότι θα πρέπει να ισοσταθμίσουμε τα συμφέροντα και τις αξίες Άρα χρειάζεται και συνέπεια. Δεν είναι μόνο το θέμα εμπορική πολιτική και των άλλων πολιτικών. Χρειάζεται συνέπεια ε, όσον αφορά και το ότι όχι μόνο η εμπορική πολιτική αλλά και άλλε πολιτικέ μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και αυτό είναι το ίδιο σημαντικό με το προηγούμενο, αν όχι πιο σημαντικό. Όπω δε προείπα, η ατζέντα διαπραγματεύσεων θα είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για την εμπορική πολιτική. Επίση όμω, θα πρέπει να βαθμίζουμε τι προσπάθειέ μα να δούμε το πώς όσα διαπραγματευτούμε θα τα τηρήσουν οι συνομιλητές μας. Άρα θα προσπαθήσουμε περισσότερο όσον αφορά τις ε, διεθνείς συνθήκες, την εφαρμογή τους, πώς θα μπορέσουμε να επενδύσουμε στις ε, αγορές των τρίτων χωρών, να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε ε, περισσότερη συμμετοχή στις προμήθειες, στους διαγωνισμούς, ούτως ώστε οι αναδυόμενες οικονομίες να είναι ανοιχτές για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, όπως κάνουμε εμείς για εκείνου στην αγορά μας, στι δικές του εταιρείε. Επίσης χρειάζεται να προσπαθήσουμε περισσότερο όσον αφορά το να συμμορφωθούν οι τρίτες χώρες με τις κρατικές, για τις κρατικές ενισχύσεις που δίνουν. Θα πρέπει επομένω να υπάρξουν περισσότερες ευκαιρίες για απασχόληση και ανάπτυξη όσον αφορά όλο τον κόσμο, ιδίως τις αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης Έχουμε μια ανακοίνωση που λέμε τις λεπτομέρειες του πώς θα αναπτυχθεί αυτή η πολιτική αργότερα. Επομένω, ο Αντώνιο Ταγιάννη, ο συνάδελφος και ο Μισελ ο συνάδελφός μου στην Κομισιόν, τώρα εκπονούμε μια καινούργια βιομηχανική πολιτική και πολιτική εσωτερική, εμπορική. Άρα θα πρέπει όλες αυτές οι πολιτικές να έχουν μεταξύ τους μια συνέπεια και έτσι όλες μαζί να συναποτελούν την εξωτερική οικονομική μας πολιτική. Στόχος μας για αυτή την ε, ανακοίνωση είναι να υπάρξει, να εκδοθεί περί τα τέλη Οκτωβρίου ε, για την εμπορική πολιτική. Όμως, θέλω εσείς κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, να μας πείτε πού πάσχει, πού έχει κενά αυτή η πολιτική, με ποιους τρόπους μπορούμε να τη βελτιώσουμε, να την κάνουμε πιο προσαρμοστική, ε, να, για να αλλάξει η ρότα της ιστορίας της πορεία του εμπορίου και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την άποψή σας στην οποία ε, στηρίζομαι πολύ. Πρόεδρος. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ξεκινούμε τη συζήτηση για τις ερωταπαντήσεις από τα μέλη της Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα θα δώσω το λόγο στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων ξεκινώντας προφανώς με το ΕΛΚ. Εάν θέλετε να ξεκινήσετε. Επίτροπε, με συγχωρείτε που καθυστέρησα. Σήμερα ήδη τέρος, αλλά είναι μια παράξενη μέρα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα θέματα. Καταρχήν, όταν μιλάμε για μια νέα στρατηγική, καταρχήν πρέπει να δούμε τι έχει γίνει και τι επιτύχαμε με την προηγούμενη στρατηγική εξωτερικού εμπορίου. Κατά την τελευταία περίοδο ήμουν εισηγητής επί του θέματος και διαπιστώνω ότι σε πάρα πολλοί τομεί δεν ήμασταν και τόσο επιτυχείς. Σκέφτομαι ε, ότι όλοι ε, ε, παραπονούνται δεν προχώρησε το θέμα του ΠΟΕ αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί και ο γύρος της ΔΟΧΑ. και εδώ δεν αναφέρουμε στο ότι υπάρχει στο τραπέζι τώρα αλλά το θέμα που πρέπει να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας και το οποίο ε, πρέπει να προχωρήσει. Όταν λοιπόν σκέφτομαι αυτά τα θέματα τότε αυτό που θα ήθελα είναι να σκεφτούμε περισσότερο πώς ε, θα διαπραγματευόμαστε για ελεύθερο εμπόριο, πού έχουμε επιθετικά συμφέροντα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Επίσης θέματα στα οποία δεν είμαστε έτοιμοι να ε, εγκαταλείψουμε τις προσπάθειες και σε άλλα όπου σε έναν κόσμο που αλλάζει πρέπει ε, να τοποθετηθούμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε με την Ινδία και οι Ινδοί είπαν ότι θα ήθελαν μια εξαιρετική μεταχείριση. Μπορούμε να προβλέψουμε εξαιρετικές ρυθμίσεις αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι για το εμπορικό, ε, την εμπορική συμφωνία ε, όλες οι εξαιρέσεις τις οποίες θα συνενέσουμε να έχουν μια συγκεκριμένη προθεσμία και ημερομηνία όπου θα εκπνεύσουν ε, μία ημερομηνία την οποία θα λάβουμε υπόψη είτε ημερολογιακά είτε βάσει ορισμένων ε, κριτηρίων τα οποία θα ε, επιδεικνύουν μία πρόοδο διότι σε όλες τις αναδυόμενες αγορές στην Κίνα, στη Βραζιλία, στην Ινδία σε όλες αυτές τις χώρες πρέπει να προβλέψουμε ότι δεν πρόκειται για στατικές εξελίξεις, για στατικές συμφωνίες, αλλά θα υπάρχει μια συνεχής εξέλιξη και δεν θα περιοριστούμε σε αυτές τις χώρες. Επίσης τα θέματα τα οποία δίνουμε τώρα δωρεάν και σκέφτομαι ε, το σύστημα προτιμήσεων, το θέμα με τους οπλισμούς, ε, όλα αυτά είναι ένα θέμα το οποίο με απασχολεί. Ε, πώς θα τα καταφέρουμε να διεκπαιρεώσουμε τα θέματα αυτά στα επόμενα έτη. Θα μπορέσουμε να τα επεξεργαστούμε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι χώρες σαν την Ινδία δεν θα μπορέσουν να αποχωρήσουν και να πούν ότι τώρα με το σύστημα των προτιμήσεων όλα αυτά τα έχουμε ήδη. Οπότε γιατί πρέπει να τα συζητήσουμε ε, σε μία συμφωνία προτιμήσεως. Επίσης ε, όταν καταρτίζεται το σύστημα των προτιμήσεων θα πρέπει να ε, διαπιστώσουμε διαπιστώσουμε ε, πώς θα προχωρήσουμε. Δηλαδή να μην υπάρχουν ορισμένοι που θα εκμεταλλεύονται. Παραδείγματο χάρη ε, τα κράτη του ε, αραβικού κόλπου πάντοτε χαίρουν ορισμένων προτιμήσεων. Είναι λοιπόν μια στρατηγική την οποία πρέπει να αναθεωρήσουμε. Αυτό που θα ήθελα είναι ότι στο μέλλον να μπορούμε να ε, ε, συνδυάζουμε καλύτερα την εμπορική πολιτική ε, με των εξωτερικών σχέσεων. Είναι μια συζήτηση την οποία κάνουμε εδώ και πολύ καιρό. Αυτό λοιπόν που με απασχολεί είναι πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους άλλους τομείς της πολιτικής για να βελτιώσουμε την πολιτική εξωτερικού εμπορίου. Παραδείγματος χάνει όσον αφορά τις πρώτες ύλες, τις συμφωνίες τις οποίες είχε συνάψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχαμε κρίνει σε μία έκθεση προ δύο ετών ε, πόσες φορές έρχεται ε, η ε, πολιτική περιβάλλοντος ή αναπτύξεως και μας λέγουν ότι θα πρέπει να στηρίξετε αυτά τα θέματα στις επόμενες συμφωνίες για εξωτερικό εμπόριο. Είναι λοιπόν διάφορα θέματα σε διάφορους τομείς ενεργειακό, γειτονίας, περιβάλλοντος Ευχαριστώ το, πολλοί τους οποίους θα έπρεπε να ε, συνυπολογίσουμε όταν συζητάμε για εξωτερικό εμπόριο. Ε, εάν μπορούσατε μάλιστα να μας δώσετε και ένα γραπτό κείμενο κατά τρόπον ώστε τύπος ε, να μπορέσουμε να σας στείλουμε τα σχόλιά μας υπό μορφή επικεφαλίδων. Θα ήθελα άλλωστε να λάβετε υπόψη σας πώς έχει αναβαθμιστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Έχω και άλλες πολλές ερωτήσεις, δεν θέλω όμως να υπερβώ το χρόνο μου και γι' αυτό θα περιοριστώ σε αυτά τα θέματα που έθιξα. Και τώρα οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες. Ο κύριος Μάρτιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα, συμφωνήσω με τον κύριο Κασπάρη ότι ο στόχος να φτιάξουμε μια ενωμένη Ευρώπη και για την εμπορική μας πολιτική με το γύρο της Δόχα φαίνεται να αποτύχαμε. Όμως οι διαπραγματευτικοί μας εταίροι, οι Αμερικανοί, η Βραζιλία και η Ινδία, στον ανανεωμένο γύρο της Δόχα φαίνεται να έχουν περισσότερες ευθύνες για την αποτυχία του πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Τώρα για τι ε, συμφωνίε μα ελεύθερων συναλλαγών. Εδώ νομίζω ότι σωστά ακολουθούμε αυτή την πορεία, αυτή την επιδίωξη. όμω, μια στρατηγική καλό είναι να υπάρχει. Να δούμε ποιε είναι οι περιοχέ, οι περιφέρειες με τι οποίε θέλουμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσει. Θα ήθελα λοιπόν να θυμίσω ότι πριν ε, θεσπιστεί αυτή η επιτροπή εντό του Κοινοβουλίου είχαμε επιτροπή βιομηχανία και εμπορίου. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τους βιομηχανικούς μας στόχους ως κοινότητας και τους εμπορικούς. Δεν νομίζω ότι κάποιες χώρες πρέπει να θεωρούν ούτως ή άλλως ότι θα κερδίζουμε πάντοτε στις διαπραγματεύσεις. Όμως να, να σκεφτούμε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ποιες ε, βιομηχανίες θεωρούμε πρωτίστη σημασία στην Ευρώπη. Ποια συμφέροντα θέλουμε να καλύψουμε πάνω απ' όλα και έτσι να διαλέξουμε τις χώρες με τις οποίες θέλουμε να ε, διαπραγματευτούμε όχι μόνο με από ποιε θα αποσπάσουμε τα περισσότερα ωφέλη και συμφέροντα, αλλά ποιε θα είναι πιο ωφέλιμες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Επίσης να πω ότι η κυρία Άστον ήταν στην Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα και είπε για την εξωτερική μας πολιτική ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να είναι ένα στοιχείο το οποίο να διατρέχει όλο το σχεδιασμό πολιτικών μας, ακόμα και την εμπορική. Αυτό βέβαια με κάνει να αναρωτιέμαι εάν εάν έχει νόημα να διαπραγματευόμαστε ρήτρε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά και τα υπεραβολοντικά στοιχεία στι ε, συμφωνίε ελευθέρων συναλλαγών. Και βεβαίω θέλουμε να προωθούνται και να συμφωνούνται τέτοιε ρήτρε, αλλά το θέμα είναι κατά πόσον είναι εφικτό. Και έπειτα ένα τρίτο ερώτημα για το ελεύθερο εμπόριο στο προηγούμενο κοινοβούλιο, στην προηγούμενη επιτροπή για το δίκαιο εμπόριο, πρέπει να δούμε κατά πόσον θα αλλάξει αυτό που γινόταν παλιότερο ότι κάθε Γενική Διεύθυνση σχεδιάζεται τη δική της πολιτική. Θα πρέπει κάποιος να αναλάβει να είναι συντονιστής των ε, πολιτικών δικαίου εμπορίου. Εσεί θα μπορούσατε να αναλάβετε ένα τέτοιο ρόλο εντό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να διασφαλίσετε το δίκαιο εμπόριο, το fair trade δηλαδή, που είναι ένα στόχος ε, που αξίζει τον κόπο, να ενσωματωθεί στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Ευχαριστούμε. Εκ των Φιλελευθέρων, ο κύριος Ρινάλντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε, για την ομιλία σας για τις αδρές γραμμές ανάπτυξης της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης. Πρέπει εδώ νομίζω να λάβουμε υπόψη και άλλες δύο παράλληλες συζητήσεις. Συζητήσεις που εξελίσσονται και στο Ευρωκοινοβούλιο τους τελευταίους μήνες και εκτός Κοινοβουλίου. Η μία αφορά την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τη θέση σε ίσια και τις συνθήκες της Λισαβόνας και έπειτα ποια είναι τα μέσα της εξωτερικής πολιτικής που θα χρησιμοποιήσουμε ως συνέπεια τη εφαρμογή τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Πρόκειται για δύο συζητήσει αρκετά δυσχερεί. Πρέπει να δούμε ποια είναι τα μέσα που διαθέτει ο, η υπατή εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική. Εξετάζοντα τα όμω, αντιλαμβανόμαστε ότι πραγματικά για την εξωτερική πολιτική τα μέσα που διαθέτουμε είναι να πιέσουμε μέσω της πολιτικής αυτής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν μας δίνει και πολλά προνόμια αλλά και σοβαρά πλεονεκτήματα. Η εμπορική λοιπόν πολιτική είναι μια σοβαρή πτυχή που καθορίζει την εξωτερική εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον εξωτερικό κόσμο. Και από την πλευρά των επιτρόπων και από την πλευρά της υπατή εκπροσώπου. Τώρα τρει ερωτήσει. Με ποιο τρόπο βλέπετε εσεί τις σχέσεις συνεργασία, τι ισορροπίες με το κολέγιο των επιτρόπων ποιοι είναι οι τομεί όπου μπορεί να υπάρχει σύγκληση και συμφωνία και ποιοι είναι οι τομεί όπου το εμπόριο προχωρά μόνο του χωρί να υπάρχει ανάγκη διαβουλεύσεων, χωρί να υπάρχει ανάγκη συνδυασμού με την αναπτυξιακή πολιτική και τι προτεραιότητε τη ύπαρξη εκπροσώπου. Και αναφέρετε κι εσεί ε, κάποια στοιχεία, φαντάζομαι, στου συναδέλφου σα. Υπάρχουν σχέσει ισορροπία μεταξύ των επιτρόπων. Έπειτα για την εμπορική μα πολιτική και την αναπτυξιακή πολιτική σε διάφορες περιφέρειες του κόσμου για τις τροποποιήσεις των διάφορων κανονισμών. Τι θα γίνει με τις χώρες ε, ΑΚΕ και την, ε, συγκεκριμένα την Σρι Λάγκα. Εδώ έχει ληφθεί μια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι μια απόφαση που θα εγκριθεί, νομίζω θα οριστικοποιηθεί μάλιστα η τελευταία αποτίμηση τον Ιούλιο Ξέρετε ότι εμείς έχουμε κάποιους ενδιασμούς για τις επιπτώσεις κάποιων, της ενισχυμένης συμφωνίας με τη Σρι Βρίσκουμε ότι εδώ υπάρχουν σφάλματα και ίσως να πληρώσουμε και ένα πολύ σοβαρό πολιτικό τίμημα. Και έπειτα και το Ισραήλ με την Παλαιστίνη. Ποια είναι τα εμπορικά μέσα για να υποχρεώσουμε να ακουστεί η δική μας άποψη, η δική μας φωνή. Ίσως να μην είναι πολλά, αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποια εμπορικά μέσα. Εσείς αναφέρατε την πρόσβαση που έχουν τα παλαιστινιακά προϊόντα. Υπάρχουν επίσης άλλες σημαντικές αποφάσεις, όπως να παγώσουμε προς στιγμή τις σχέσεις μας με το προσάρτημα της Συμφωνίας Συνεργασίας με το Ισραήλ. Όμως, ποιες είναι οι διάφορες μορφές της εμπορικής πολιτικής μπορεί να χρησιμοποιηθούν από το φως και των πρόσφατων γεγονότων για να ασκήσουμε πίεση στην περιοχή αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Μετά τις πολιτικές ομάδες, μάλλον τις πολιτικές ομάδες καλό είναι να τις χωρίσουμε σε δύο ομάδες ερωτήσεων, ώστε να μπορέσει ο Επίτροπος να απαντήσει χρονικά πιο κοντά στις ερωτήσεις που τέθηκαν. Ο κύριος Λάντο λοιπόν και μετά ο Επίτροπος για μια σύντομη απάντηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι άπαξ και αναπτύσσουμε μια νέα στρατηγική, όπως το είπατε και εσείς κύριε Επίτροπε, πρέπει να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και τι απολογισμό μπορούμε να κάνουμε της προηγουμένης στρατηγικής. Ε, στα τρία χρόνια αυτά είχαμε πρώτα μία διατροφική κρίση η οποία ήταν συνδυασμένη με μία κρίση στις αγορές των ε, γεωργικών ε, προϊόντων, μία ενεργειακή, μία κοινωνική, μία περιβαλλοντολογική και οικονομική κρίση και στην τελευταία φάση η δημοσιονομική πολιτική ήταν πάρα πολύ ενεργή με επιδοτήσεις σε ορισμένους τομείς ή με παρεμβάσεις στον οικονομικό τομέα των κρατών. Δηλαδή βλέπουμε τελευταίως ε, πόσο δραστηριοποιούνται ε, οι υπεύθυνοι των εξαγωγικών ε, επιδοτήσεων για να στηρίξουν τις ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες και για να ε, επέμβουν βραχυπρόθεσμα. Στις δημόσιες όμως συζητήσεις εφόλης της ύλη, όταν μιλάμε για ολοκλήρωση μιλάμε για ντάμπινγκ κοινωνικό, φορολογικό, νομισματικό και ακόμη και εδώ δεν, καταφέρνουμε σήμερα να ερμηνεύσουμε επαρκώς τα θέματα αυτά σε μία πολιτική, οικονομική ή κοινωνική. Θέλω λοιπόν να επιμείνω στο εξής τι είναι ο απολογισμός εμπορικά των κρίσεων που διεξήχθησαν τα τελευταία χρόνια. Ξέρω ότι όλοι ξέρουμε ότι το εμπόριο μπορεί να μας βοηθήσει να εξέλθουμε από την κρίση αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε αξιολογήσει επαρκώς κατά ποιον τρόπο η απελευθέρωση του ε, εμπορίου ίσως επιδίνωσε ή επιτάχυνε την κρίση. Παραδείγματο χάρη η απελευθέρωση των οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών τα τελευταία τελευταία χρόνια ε, οδήγησε στην κρίση τα τελευταία δύο χρόνια ή τους τελευταίους 18 μήνες μετά την, ε, από αυτό είναι βασικό ότι πάντοτε σκεφτόμαστε στις διαρθρωτικές ευρωπαϊκές ε, πολιτικές ως πολιτικές οι οποίες επιτρέπουν να προσαρμοστούμε στην ε, ε, παγκοσμιοποίηση. Θυμάμαι ε, για, στην απελευθέρωση των αλλιευτικών υπηρεσιών όπου μου εξηγούσαν ότι αυτό επιτρέπει εις την Ευρωπαϊκή Αλία να προσαρμοστεί στην παγκοσμιοποίηση της αλίας και τελικά έχουμε κατά λάθο ε, μία, βιομηχανική ε, πολιτική στην Ευρώπη διότι ανοίγουμε έναν τομέα, αναπτύσσουμε έναν άλλον χωρίς όμως να υπάρχει μία προφανής ε, εξέλιξη της βιομηχανικής πολιτικής. Λοιπόν, στην Τόχα αυτό έχουν σταματήσει συζητήσεις. Ποια πρέπει να είναι η αναδιάρθρωση της στρατηγικής της Ευρώπης για να ξεκινήσουν και πάλι συζητήσεις. Όσον αφορά τις διημερείς συμφωνίες χωρώνα και ή άλλων, κατά πόσον ε, τα ε, κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούμε μπορούν να συμβάλλουν ώστε οι συζητήσεις να βασίζονται σε κριτήρια τα οποία ενδιαφέρουν την Ευρώπη. Τρίτον, πώς μπορούμε στην οικονομική πολιτική σήμερα να προσθέσουμε τις ε, προκλήσεις και είμαστε σε 500 δισεκατομμύρια ε, ευρώ για επιδοτήσεις. Οπότε πώς εξηγούμε τόσο τεράστιες και απαράδεκτες επιδοτήσεις σε τομείς όπως ο ενεργειακός. Τέλος, έχετε δεσμευτεί και είμαστε ευτυχείς ε, για τα θέματα της Κορέας προτού εφαρμοστεί ο μηχανισμός που έχει αποφασιστεί πώς πρέπει να λειτουργήσουμε ώστε η ανανέωση των διαπραγματεύσεων με το Μερκοσούρ να μην παρουσιάσει τα ίδια προβλήματα διότι εσείς είσαστε αρμόδιος αλλά πιστεύω ότι στα θέματά σας θα έπρεπε να έχετε μία συζήτηση με το Κοινοβούλιο. Κύριε Επίτροπε, θέλετε να απαντήσετε στις τέσσερις πρώτες ερωτήσεις. Ναι, κύριε Πρόεδρε, στα γαλλικά κατάλαβα. Από ό,τι κατάλαβα ότι αυτό το οποίο θέλουμε είναι να μου υποβληθούν οι ερωτήσεις, να τις λάβω υπόψη και κατόπιν τις ιδέες σας να τις εντάξω ή στην αναγύρωση που εκπονούμε. Αλλά φυσικά δεν έχω πρόβλημα να απαντήσω στις ε, συγκεκριμένες ερωτήσεις. για αυτό που ερωτήθηκε στον αυτό το Μερκοσούρα, ε, Νίκ Ζαντό, στο Σώμα των Επιτρόπων είπαμε ότι θέλουμε να δώσουμε νέα όθηση στις διαπραγματεύσεις και την ίδια μέρα την επομένη ήρθα και τα είπαμε εδώ. Και το Συμβούλιο είπε ότι προχωρήσατε χωρίς να μας δείξετε τη γνώμη και εκ των υστέρων μόνο μας ενημερώσατε μια, δυο μέρες μετά στην Trade Policy Committee. Το δε πλεονέκτησε σε συγκεκριμένη περίπτωση όσον αφορά το Συμβούλιο, την ενημέρωση. Αλλά βέβαια και το Κοινοβούλιο αισθάνθηκε προσβολημένο και υπήρχαν επίση και κάποιε χώρε μέλη που είπαν ότι δεν συμφωνούμε γιατί θα έπρεπε να έχει προηγηθεί κάποια διαβούλευση. Εγώ είπα ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα να συζητήσω με τους πάντες και να λάβω υπόψη τις αρμοδιότητες του κάθε θεσμικού οργάνου. Και εσείς επίσης τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι υπάρχει εντολή διαπραγματευτική για το Μερκοσούρ. Εντολή σαφή. Οπότε και εμεί ξεκινήσαμε και πάλι τι διαπραγματεύσει στα πλαίσια τη εντολή αυτή. Μια που εμπίπτει στι αρμοδιότητέ μα. Βεβαίω και πρέπει να ενημερωθεί το Κοινοβούλιο, το συζητήσουμε. Βεβαίω και σεβόμεθα τι δικέ αρμοδιότητε, αλλά και εμεί έχουμε τι δικέ μα. Καλύτερο τρόπο λειτουργία αυτού του θεσμικού τριγώνου είναι το να σέβεται ένα αρμοδιότητε του άλλου. Α, δεν ήταν ζωντό. Άρα, σεβασμός της κατανομής της διαίρεσης των αρμοδιοτήτων. Αυτό, αυτό χτίζει καλύτερες φιλίες. Τώρα, όσον αφορά το dumping. Πιστεύετε ότι η απορρίθμιση στα χρηματοπιστωτικά δεν είναι η μόνη αιτία της κρίσης. Οπότε, τελικά είναι θέμα πεπιθήσεων. Θεωρώ πάντως ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ήταν μια από της κρίσης κρίση, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι η απορρίθμιση έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον, θα μας οδηγήσει σε κάποια αλλαγή της φύσης των ιδρυμάτων αυτών που έχουν αποκτήσει θεσμικό ρόλο. Και κάποιες ε, εταιρείε κάποια νομικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει πρόσβαση στις επιχειρηματικέ δραστηριότητε σε βιομηχανία, στην οικονομία, στην κοινωνία πρωταγωνιστικά πρόκειται για μια βιομηχανία τραπεζικών προϊόντων Επομένω, έχει αλλάξει η φύση αυτών των ιδρυμάτων για πολλούς λόγους Και βέβαια δεν ξέρω αν είναι θέμα δικό σας δικής αρμοδιότητας αυτής εδώ της Επιτροπής, αλλά η πρώτη και η δεύτερη συνδίκη της Βασιλείας και κυρίως η δεύτερη κυρίως η δεύτερη έχουν οδηγήσει στην αξιοποίηση των τραπεζικών προϊόντων οπότε και έτσι οδηγηθήκαμε στο τόσο ευμετάβολο της αγοράς φτάνει σε τρομερά επίπεδα. Και αυτό βεβαίω βοήθησε στο να υπάρχουν ε, ανισορροπίε στι ε, αγορέ. Επομένω δεν είναι θέμα απορρίθμιση. Το θέμα ήταν, ήταν κατά τη γνώμη μου, το ότι έγινε ρύθμιση λανθασμένη. Αυτό το περίφημο market to market. Έτσι είχαμε την εκτροπή. Το πώς δούλεψε δηλαδή αυτό το σχήμα και αυτό δεν πάει να πει όμως ότι δεν υπήρχε ρύθμιση. Όχι, όχι, όχι, ήταν πράξεις που γινόντουσαν νόμιμα, διότι δεν υπήρχε κάλυψη νομική αρκετή. Ή πάλι ότι αυτό όλα μας ήταν ξένα και, στο, και στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο και, και σε εσάς. Δεν φταίει το ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι η αιτία και οπότε φταίει γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να κάνει την απορρίθμιση. Θα πρέπει αυτό να μου το αποδείξετε. Από πού και ως πού. Από πού και ω πού είναι θέμα απορρίθμιση. Το κάτι το οποίο δεν γίνεται εύκολα. Bon, comment euh, euh? Πάμε επομένως τώρα για τι διαμετεύσεις για την Ντόχα. Ούτε νομίζω ότι είναι θέμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει καινούργια όθηση και να επαναρχίσει τι σχετικέ διαπραγματεύσει, διότι είχαμε αυτή τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Γενέβη το 2008, τον Ιούλιο. Ιούνιο. Και είχαμε κατόπιν αυτή την αντιπαράθεση με Ινδία και με ΙΠΑ. Οπότε η υπόθεση δεν προχώρησε. Θεωρώ δε ότι Ισχύει πως τον Ιούλιο του 2008 στη Γενέβη αυτό το οποίο ήταν το διακύβευμα δεν έλαβε μορφή συμφωνίας γιατί θα πρέπει τώρα να υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Όμως, αυτό το είπα και στους Αμερικανούς φίλους, ότι θα πρέπει και αυτοί να δουν από τη δική τους πλευρά να, δουν, να ψάξουν τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει ούτως ώστε να καταστεί εφικτό να απεμπλακεί η κατάσταση. Δεν νομίζω ότι ε, συμφέρον και ενδιαφέρον την Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνει αυτό. Αυτό το οποίο τότε διακυβευόταν το 2008 ήταν μια συμφωνία που θα ήταν για μας αποδεκτή. Βέβαια, δεν θα ωφελούνται και τα δύο μέρη το ίδιο. Εντάξει, εμεί έχουμε ανοιχτή στάση. Είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε. Να ξεκινήσουμε όμως εμείς, εμείς πώς με νέες παραχωρήσεις στη Γεωργία, για παράδειγμα. Ε, δεν νομίζω ότι αυτό θα σας αρέσει. Με λέτε να, να λάβουμε την πρωτοβουλία και να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις. έτσι και το κάνω αυτό ελίμονό μου. Στην κοιλωτίνα. Ναι, να κάνουμε θυσίες για την Ευρώπη, αλλά μην το παρακάνουμε κιόλα. Μην το παρακάνουμε. Uh, oui, dans free trade agreements. Free trade agreements, συμφωνίες ελευθερών εμπορίου. Par exemple, donc, est επειδή μιλάμε για τα κριτήρια βιωσιμότητας, νομίζω ότι εν μέρει αυτό γίνεται. Όμως, πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Προσεγγίζουμε κάποιες αγορές ανάλογα με το τι θεωρούμε ότι είναι σημαντικό τομέα για την βιομηχανική μας πολιτική. Πρέπει όμως να προσεγγίζουμε αγορές όπου υπάρχει και κάποια αγοραστική δύναμη. Μπορούμε βεβαίω να αναμένουμε, να προσδοκούμε εξελίξεις. Αλλά αυτό μας ζητάτε και από τη στρατηγική 2020. Αναζητούμε αγορές για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Euh, euh, euh, Έτσι λοιπόν η βιωσιμότητα με τις οριζόντιες κοινωνικές ρήτρες είναι κάτι που λαμβάνουμε υπόψη. Όμως Πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις προτεραιότητε τη βιομηχανικής μας πολιτικής. Και το θέμα είναι ποιο αποφασίζει ποιοι είναι αυτοί οι τομείς. Είναι οι κυβερνήσει. Οι κυβερνήσει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι έχω την τάση να πιστεύω ότι οι οικονομικοί φορείς, οι βιομηχανίες, οι εταιρείε. δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να είναι οι ίδιοι που θα μας πούν τι πρέπει να εντοπίσουμε στο τομέα προτεραιότητας. Εάν ο ίδιος ο χώρος δηλαδή της οικονομίας θα πρέπει να μας πει που να επικεντρωθούμε. Qui στην Ευρώπη λοιπόν το τι λειτουργεί καλύτερα, ίσως είναι κάπως τυχαίο, αλλά είναι μια, μια επιλογή που έχει γίνει από την ίδια την αγορά, την οικονομία. Και βεβαίως ε, και με την ε, συμμετοχή του κοινωνικού περιβάλλοντος και του χρηματοπιστωτικού. Τώρα, οι επιδοτήσεις για, τη... για τα ορυκτά κάψιμα πώς αυτό θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στην εμπορική μας πολιτική. Πράγματι, υπάρχουν σημαντικές επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα. Όμως νομίζω ότι είναι επιδοτήσεις προς μία βιομηχανία που δεν είναι φυσικά η μόνη πηγή ενέργειας. Είστε όμως πεπισμένοι κι εσείς ότι πρέπει να πάυσουν οι επιδοτήσεις για μια στιγμή. Σε μια στιγμή μάλλον θα πρέπει να σκεφτούμε πως πρέπει να προβλεφθεί και αύξηση, να δούμε λόγω χάρη την αιωλική ενέργεια. Εάν το δούμε από οικονομική άποψη, οι επιδοτήσει είναι ακόμα πιο σημαντικέ από τα αρκτικά καύσιμα. Στο βαθμό λοιπόν κατά τον οποίο οι ανάγκες της βιομηχανίας δεν αυξάνονται, πρέπει να παραμείνουμε και στη λογική των επιδοτήσεων, αλλιώς χάνουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Ε, γιατί εδώ μιλάμε για την ε, ενέργεια που είναι σημαντική. Αν λέτε για 500 εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεων στις, στα αυτό εξεπακούει και υπονοεί ότι αν υπήρχαν άλλες δυνατότητες θα μειωνόταν αυτό το ποσό. Euh, Βραχυπρόθεσμα ίσως τα ορυκτά καύσιμα παρουσιάζουν και πολλά μειονεκτήματα. πρέπει να τα δούμε διαφορετικά, διότι μετά την πυρηνική ενέργεια είναι πιο γόνιμη αγορά. Δεν άκουσα επίσης προβληματισμούς για την πυρηνική ενέργεια να εκφράζονται. Για τη Μερκοσούρ, νομίζω ότι ήδη απήντησα. Στον κύριο Μάρτιν τώρα, για εντολότερες συνεργειακές σχέσεις σχέσεις μεταξύ εμπορικής και βιομηχανικής πολιτικής ενδεχομένως να αληθεύει αυτό. Όμως θα πρέπει κανείς να σχεδιάσει την βιομηχανική πολιτική. Και βεβαίως και συζητούμε με τους ηθήνοντες της βιομηχανικής πολιτικής. Δεν είναι μόνο δικαίωμα και προνόμιο αυτό να συζητούμε με τους συναδέλφους της βιομηχανικής πολιτικής, είναι και υποχρέωση. Και πραγματικά δεν υπάρχει περίπτωση να συζητήσω με κάποιον ε, εκπρόσωπο βιομηχανικού κλάδου που να μην μου πει ότι ο δικό του βιομηχανικό κλάδο είναι στρατηγική σημασία. Αυτό δεν υπάρχει. Ε, eh, uh, um, Βεβαίω, οι άνθρωποι δεν είναι πάντοτε σε θέση να κάνουν τις σωστές επιλογές, παρόλο που τα πάντα εδώ είναι θέμα επιλογής. Τέλος πάντων, αν στι Ρητρε συμπεριλάβουμε... Αν στι συμφωνίες μάλλον συμπεριλάβουμε τις ανάλογες ρήτρες. Σαφώς και πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι ρήτρε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα με τη Σρι Λάγκα. Δεν έχω την αίσθηση όμως ότι όλα τα κρατημέλη συμφωνούν. Όμως εάν το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να κάνουμε κάποια επιλογή. Εγώ θα συμπεριλάβω πολύ αυστηρέ προποθέσει αυτέ τι συμφωνίε. Θα επιμείνω γι' αυτό. Δύσκολα θα υλοποιηθούν. Ίσως θα ήταν καλύτερα να ήταν κάπως πιο υπηκής. Πάντως αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Και ξεχωριστά οι συμφωνίες και συλλογικά. Έχω την αίσθηση ότι προσπαθούμε να είμαστε πολύ κομψοί στη διατύπωση για να ικανοποιήσουμε και τις δύο πλευρές, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε εάν μπορούν να φτάσουν στις προσδοκίες που θέτουμε και οι δύο πλευρές. Πρέπει λοιπόν να είμαστε από τη μια επίκηση, αλλά να μπορούν οι συμφωνίες και να εφαρμοστούν. Για το δίκαιο εμπόριο, το fair trade, Μου ζητήθηκε συντονισμό. Δεν μου ζητήθηκε μάλλον συντονισμό ακόμη για το θέμα αυτό, αλλά αν μου ζητηθεί δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτό ίσω θα πρέπει να γίνει σε μια ξεχωριστή συζήτηση. Τι θα γίνει δηλαδή με συγκεκριμένε χώρε στον κόσμο και ιδίω με τι ε, αναπτυσσόμενε, τι λιγότερο αναπτυγμένε μάλλον. Και το θέμα δεν είναι απλώ δασμολογικό, είναι πολύ πιο περίπλοκα εδώ τα πράγματα. Πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία εκμάθησης όχι μόνο με τα εμπορικά ζητήματα, αλλά και με το δίκαιο εμπόριο. Ζήτησα κάποια αριθμητικά στοιχεία για τα ορυκτά, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Και αν τα αφαιρέσει κανείς αυτά, δεν μένουν και πολλά. Στον κύριο Ρινάλντι, και τη σύγκριση που κάνατε μεταξύ εμπορικής και εξωτερικής πολιτικής, την αντιπαράθεση μάλλον. Ε, νομίζω, αν δει κανεί τι στήριξη μπορούμε να έχουμε στις διεθνείς μας διαπραγματεύσει όντω η εμπορική πολιτική είναι η σημαντικότερη πολιτική που διαθέτουμε. Θα έπρεπε να υπάρχει προσεκτικός συνδυασμός εξωτερικής και εμπορικής πολιτικής. Βέβαια αυτό δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα. Ένα από τα σημαντικά στοιχεία είναι ότι η κυρία Άστον αυτό το γνωρίζει πολύ καλά. Έχει ασχοληθεί με την εμπορική πολιτική για αρκετό καιρό. Όταν λοιπόν συζητήσαμε προβλήματα που υπάρχουν, είδαμε ότι έχουμε ακριβώς την ίδια στάση στα πράγματα. Για τις G, συμφωνίες GSP και GSP-SYN, Βρισκόμαστε στη φάση των διαβουλεύσεων. Και θα προχωρήσουμε σε συμφωνίες γενικές GSP μέχρι του χρόνου. Αλλά δεν θέλουμε να έχουμε αυτή τη στιγμή μια απλή μετακύληση και μια υποχρεωτική αλλαγή στον ισχύοντα κανονισμό. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε με τα μέσα των ε, εμπορικών μα συμφωνιών ε, στην περίπτωση του Ισραήλ. Κάτι μπορούμε να κάνουμε. Ήδη έχουμε ζητήσει από το Κοινοβούλιο να λάβει κάποια πρωτοβουλία. Είδαμε πρόσφατα τη συμφωνία συνεργασίας με το Ισραήλ. Επί τη ευκαιρία μάλιστα της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας τότε υποχρέωσε το κοινοβούλιο το Ισραήλ να δεχτεί την εξαγωγή προϊόντων απευθείας στην την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα λοιπόν έχουμε συμφωνήσει εντός της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τα κράτη-μέλη να είναι απαλλαγμένα από δάσμους τα προϊόντα που εξάγονται από τα Παλαιστινιακά εδάφη. Μπορούμε λοιπόν σίγουρα να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και για τους Παλαιστινίους βεβαίως θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα ακριβώς θα γίνει, γιατί αυτό θα καθορίσει και την επιλογή μας έναντι του Ισραήλ. Όμως δεν πρέπει η πίεση να είναι και υπερβολική. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει και πολιτική τόλμη ταυτόχρονα για να φτάσουμε στο τέρμα. Πάντως σίγουρα κάτι μπορεί να γίνει. Uh, για τον ε, για το γύρο της Δόχας, κύριε Κασπάρη, νομίζω ότι απάντησα. Και για τις διαπραγματευόμενες χώρες επίσης. Αληθεύει ότι αν δούμε τις συμφωνίες του Γενικού Προτιμησιακού Συστήματος <clears throat> και τις ενισχυμένες τέτοιες συμφωνίες, GSP και GSP+, σίγουρα θα πρέπει να είμαστε επιλεκτικοί και δεν θα πρέπει, όπως είπα, να γίνει μια απλή μετακύληση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη το πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση των περισσότερων χωρών με τις οποίες είχαν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις σε άλλη χρονική στιγμή. Τώρα για το έγγραφο. Υπάρχει τέτοιο έγγραφο και μπορείτε και να το συμβουλευτείτε. Μόλις όμως είναι έτοιμη και η ανακοίνωση της Επιτροπής, θα έρθω και πάλι στην Επιτροπή σας πριν τεθεί επιτάπητος προς συζήτηση η ανακοίνωση αυτή για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις μας. Σας ευχαριστούμε. Επίτροπε, χάσαμε αρκετό χρόνο, θα πρέπει να επιταχύνουμε. Διότι όχι μόνο οι πολιτικές ομάδες δεν έχουν ολοκληρώσει με τις ερωτήσεις τους, αλλά έχω και άλλα αιτήματα για το λόγο. Μην ξεχνάτε ότι ο βασικός στόχος όλης αυτής της συζήτησης είναι να δούμε τους προσανατολισμούς και τις προτεραιότητες της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ερχόμενη δεκαετία υπό το φως της στρατηγικής το 2020 για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, όπως ακριβώς ήδη εγκρίθηκε από το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Στέρντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, υποθέτω ότι αυτή τη στιγμή ασχολείστε με τους συντονιστές. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την ε, πολύ σωστή και ικανοποιητική απάντηση αλλά ε, είναι σαν να καλύψατε τα πάντα από τις χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις μέχρι την πυρηνική ενέργεια και ούτω καθεξής. Ε, είμαι υπέρ της πυρηνικής ενέργειας. Αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής Ίσως ε, έχω λάθος, αλλά είχαμε επαρκή νομοθεσία. Ίσως όχι καλή, αλλά δεν υπήρχε ε, δεν υπήρξε η ιδέουσα προσοχή στα, τοξικά δάνεια ε, και μιλώ εδώ μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε περισσότερη νομοθεσία διότι όσο περισσότερη νομοθεσία τόσο πιο δύσκολη η ασυνόμευση Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν τι νομοθεσία έχετε κατά νου από αυτή τη θέση διότι δεν θα πρέπει να καταρτήσουμε νομοθεσία η οποία θα πνίξει τις δυνατότητες ε, νέων ε, επιχειρησιακών ευκαιριών διότι είναι ο μόνος τρόπος να βελτιωθεί η Ευρώπη και να αντεπεξέλθει των χρεών της. Εγώ θα κάνω την έκθεση για την, ε, το ελεύθερο εμπόριο με την Κορέα που είναι ίσως το πρώτο θέμα στα Σπάργανα δηλαδή και θα αποτελέσει το πρότυπο και για τις συμφωνίες με τις άλλες χώρες. Οπότε εάν δούμε ότι είναι καλή η μορφή θα τη χρησιμοποιήσουμε και περαιτέρω. Όσον αφορά την Τόχα, συμφωνώ με αυτά που είπε ο Ντάνιελ. Ε, πιστεύετε πραγματικά ότι η Ντόχα θα επιβιώσει, ότι οι άνθρωποι θα επανέλθουν στο τραπέζι. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι η πιο προστατευτική χώρα στον κόσμο. Χειρότερη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη Σουηδία, παραδείγματος χάρη. Πιστεύετε λοιπόν ότι έχουμε τέτοια δυνατότητα διότι ε, θα γίνουν διμερείς και όχι πολυμερείς συμφωνίες. Αναρωτιέμαι λοιπόν εάν πιστεύετε ότι το μέλλον πηγαίνει έτσι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο εκπρόσωπος της ΓΟΕ. Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, Επίτροπο Ντεγκούχτ για την επανειλημμένη ευκαιρία που μας δίνεται να συζητήσουμε τα θέματα αυτά μαζί του και ίσως καλό θα ήταν αυτά να γίνονται όχι μόνο όταν ε, τελειώνουν ορισμένες διαβουλεύσεις αλλά να ακούει και τη δικιά μας Επιτροπή. Ε, δηλαδή πρέπει και εμείς να μπορέσουμε να σχολιάσουμε την μελλοντική εξωτερική πολιτική για να είμαστε σοβαροί. Τα θέματα λοιπόν τα οποία μας κινούν τα έχουμε λάβει υπόψη μας και ε, όσον αφορά την περαιτέρω εξέλιξη της, ε, ε, του, ΠΟΕ σαν μέρος της εμπορικής συμφωνίας όλα αυτά συζητούνται και νομίζω ότι ο Επίτροπος είναι σε δύσκολη θέση αν νομίζει ότι εμείς ψάχνουμε για γιατροσόφια αλλά όταν μιλάμε για την κατεύθυνση της εμπορικής, εξωτερικής εμπορικής πολιτικής και να συμφωνήσουμε θα πρέπει να υπάρχουν ορισμένες συμπεφωνημένες προϋποθέσεις. Παραδείγματος χάρη, στις διαβουλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν μιλάμε για την Οικονομική Επιτροπή, την Οικονομική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπου το Συμβούλιο ξεκινά από νέα δεδομένα για το πώς θα αντεπεξέλθουμε από την κρίση. Είναι κάτι το οποίο έχουν ε, σκεφτεί, ε, δηλαδή επαρκεί επαρκή με την διαδικασία και την τωρινή ζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και ε, τότε ε, ερωτάτε σχετικά με την συνεταιριστική ε, σχέση σκεφτόμαστε με τους ομολόγους μας σκεφτόμαστε την ανταγωνιστικότητα το μέλλον των ε, ε, των εργαζομένων μας ή πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει μόνο εάν οι εργαζόμενοι στην ε, Κίνα, στην Κορέα, στη Βραζιλία θα έχουν επίσης ένα επιπλέον κέρδος από αυτές τις ε, εμπορικές συμφωνίες. Οπότε η αηφορία ε, της ευρωπαϊκής της κοινωνικής πολιτικής και της οικονομικής πολιτικής είναι σημαντική. Ας πάρουμε το παράδειγμα της πετρελοκυλίδας και του ατυχήματος στον κόλπο του Μεξικού. Πόσο αυτό μας επηρεάζει για τις κοινέ σχέσεις που έχουμε ε, με τις Ηνωμένε Πολιτείε ε, αν συζητάμε για μελλοντικές σχέσεις ή με τον Καναδά. Μία, ε, μία οικολογική κατάσταση καταστροφή ή ε, την άντληση πετρελαίου πώς αυτό θα μας επηρέαζε. Ε, πρέπει λοιπόν να συζητάμε και τις εταιρικέ σχέσεις. Πρέπει να τις συζητήσουμε και στον ΠΟΕ, πρέπει να έχουμε θάρρος και να αναθεωρήσουμε το σκεπτικό μας και αν οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν επιθυμούν να θίξουν τα θέματα αυτά, εμείς πρέπει να επινοήσουμε νέες διεξόδους και να τα συζητήσουμε και τέλος, δεν θέλω να μακρηγορήσω υπερβολικά, προηγουμένως Είπατε, ε, μιλήσατε για την παγκόσμιο διακυβέρνηση επί της οποίας είπατε ότι πρέπει να συμφωνήσουμε με τις διάφορες άλλες ελεύθερες δομές. Ε, στα πλαίσια της, ε, του ΠΟΕ σε όλα τα θέματα τα οποία δημιουργούνται και αυτό θεωρούμε ότι είναι μια πολιτική εμπορική ή για την περαιτέρω πορεία. Ο κ. Ντάτμαρα το ε, ε, κόμματος συντηρητικών. Καταρχήν ε, θέλω να συγχαρώ τον Επίτροπο για την πολύ σαφή παρουσίαση του και να του πω ότι είστε πολύ καλύτερος από τον προκάτοχό σας ο οποίος ε, παρόλα αυτά ή προκάτοχό σας προήχθη στο θέση της υπάτου εκπροσώπου παρόλο την τραγική παρουσίαση εδώ. Ο Ντέβιντ Μάρτιν παρόλη την ευγλωτία του και το ε, γοητεία του αναφέρθηκε στα ανθρώπινα δικαιώματα και όλοι είμαστε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά αυτό σημαίνει για όλους αυτό που θέλουμε να σημαίνει και αυτό που δεν ξέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ξέρει ο Ντέβιτ Μάρτιν είναι ότι εις, ε, την Αγγλία αυτό έχει ερμηνευθεί από τα δικαστήρια ε, σαν ε, μία χάρτα για τους απατεώνες. Οπότε, όπως είπε προηγουμένως ο κύριος Ρινάλντι που έφυγε, η Σριλάνκα που είναι μέλος της, ήταν μέλος της κοινοπολιτείας έχει τιμωρηθεί και πιστεύουμε ότι έχει τιμωρηθεί αδίκως εν ονόματι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον Επίτροπο εάν είναι δυνατόν να μου διευκρινίσει ποια είναι τα προγράμματα του Επιτρόπου και των συναδέλφων του στο τμήμα εμπορίου ε, για να επιστρέψει στη Σρι Λάγκα το σύστημα ή προτίθενται ε, άλλες χώρες όπως και η Σρι Λάγκα να τιμωρηθούν ε, επί της ιδίας υποκειμενικής βάσεως και τέλος θα ήθελα να πω στον Επίτροπο ότι το εμπόριο του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων χωρών θα ε, ε, παρεμποδιστεί από τις πολιτικές επιταγές άλλων κρατών και θα ήθελα να ακούσω με μεγάλο ενδιαφέρον τα σχόλιά του. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι θα ήταν ε, ε, ε, θα, πρέπει να δώσω το λόγο και στους εκπροσώπους της Επιτροπής Αναπτύξεως που μου έχουν ζητήσει να λάβουν το λόγο. Ο κύριος Ντέβα λοιπόν. Ευχαριστώ. Πάντοτε είναι χαρά μου να ε, ε, ε, συζητάμε με τους συναδέλφους και χαιρετίζω και τον Επίτροπο. Εδώ εκπροσωπώ την Επιτροπή Περιβάλλοντος και τον Πρόεδρό της και χαιρετίζουμε τις δημόσιες διαβολεύσεις που έχει ξεκινήσει ο Επίτροπος και σύμφωνα με ε, την συνθήκη της πρέπει να ε, μειώσουμε την φτώχεια και να βελτιώσουμε τις αναπτυξιακές μας πολιτικές. Για αυτούς τους λόγους υπάρχουν ορισμένες ανησυχίες στην, στην ε, Επιτροπή μας ότι οι δημόσιες διαβουλεύσεις έχουν εμφανιστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε τα αποτελέσματα ε, να μην ε, ε, είναι διάφανα και το αποτέλεσμα είναι να ξέρουμε ποιος έχει πει τι και ποιες ήταν οι ανησυχίες του καθενός για να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε στη συζήτηση. Και τώρα ξαναδίνουμε τον λόγο στον κύριο Επίτροπο για να απαντήσει αυτόν τον δεύτερο γύρο των ερωτήσεων. Και άλλοι συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Θα τους δώσω το λόγο για έναν τρίτο γύρο των απαντήσεων. Πρώτα πρώτα αυτό που ρώτησε ο κύριος στάδιο. Ξέρουμε ότι ετοιμάζεται κάποιους ε, κανονισμούς για τα χρηματοπιστωτικά. Ξέρετε ότι δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Εγώ απλώς έκανα ε, μια γενική τοποθέτηση για την κρίση. Να δεν πάμε τώρα στις λεπτομέρειες. Τώρα, με την Κορέα τι γίνεται. Μιλούμε για μια συμφωνία ελευθερών εμπορίου αλλά δεν έχουν όλοι μας οι εταίροι το ίδιο επίπεδο ανάπτυξης όπως η Νότια Κορέα. Οπότε, ανάλογα με την ανάπτυξη, απευθύνεται κανείς και σε κάποιον. Και για την επίλυση των διαφορών. Νομίζω ότι είναι η σχετική συμφωνία πάρα πολύ αξιόλογη. Αυτό το λέω με σιγουριά. Επί του παρόντος πάντως θα συνεχίσουμε τις διμέρειες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Πάντως είμαι πεπισμένος ότι αργά γρήγορα θα υπάρξει συμφωνία για την Τόχα. Δεν νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να θίγονται σημερινά μπορούν να συνεχίσουν να αυτή τη στάση ε, νομίζω του χρόνου που θα φτάσει στο μισό η θητεία του Πρόεδρου κάτι θα γίνει κάποια θετική εξέλιξη θα έχουμε αναθεώρηση των μέσων οικονομικής πολιτικής, εμπορική πολιτική αφορά εταιρικέ σχέσεις βεβαίως. Να κοιτάξετε και την συμφωνία με την Κορέα. Είμαστε σε επαφές με την Ινδία για ατομικά και συλλογικά εργατικά δικαιώματα αλλά κανείς δεν τα βλέπει τα πράγματα έτσι όπως εμείς αλλά έχετε δίκιο. Είναι και θέμα του τι ρόλο θέλει να αναλάβει έκαστος σε αυτόν τον κόσμο. Τι άλλα θέματα που να σε μια εμπορική συμφωνία. Μίλησατε και για τον κόλπο του Μεξικού. Δεν είμαι ειδικό να μπω στι λεπτομέρειε, αλλά σίγουρα πρόκειται περί ατυχήματο. και βέβαια αφορά τα τα ύδατα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τις κακές εξελίξεις. Κάνουμε ό,τι μπορούμε από πλευρά διαχείρισης, εγκαταστάσεων, πλατφόρμες θαλάσσιες, άλλη άλλοι είναι αρμόδιοι γι' αυτό, άλλη επιτροπή. Και ξεκινώ από αυτό πραγματικά για το οποίο πραγματικά ήταν τραγικό. Βεβαίω και πρόκειται να συζητηθεί αυτό για πολύ καιρό, αλλά πάντως νομίζω το ίδιο ισχύει και με αυτό που στον Καναδά. Είναι βέβαια και θέμα οικονομικό με όλο αυτό το φυσικό που βρήκανε κοντά στην φαίνη του εδάφους. Δεν ξέρω. Θα δούμε, θα δούμε. Τέλος πάντων. Δε, αυτά τώρα δεν είναι τα δικά μας θέματα, Πρόεδρε. Έχουμε ένα σωρό ερωτήσεις για όλα τα θέματα, εφόλης της ύλης εδώ. Μια πέστη μας τώρα. Προσπαθούμε, ναι, να δούμε τι, τι τους στο, G20, τι τους διακυβέρνηση παγκοσμίου μπορεί να γίνει. Βέβαια το G20 είναι G20, δεν είναι ε, εκεί οι εξελίξεις, είναι πολυμερής ε, οργανισμός και εδώ υπάρχει ενδιαφέρον θέμα για το, για το κοινοβούλιο. Ο ΠΟΕ, ο ΚΤΑΔ, όλοι αυτοί οι φορείς μπορούν να κάνουν πολλά. Φυσικά και είναι πάρα πολύ θετικό το ότι το G20 μπορεί να δώσει κάποια όθηση αλλά αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να έχουν κάθε εντολή οι και με αυτή την εντολή να προχωρήσουν όμως ξαφνικά πώς, πώς να προκύψει λύση από το G20. Καθένα άλλο βλέπει τα πράγματα. Μπορεί να ξεκινήσει μια νέα διαδρομή τριετής. Να. Έχουν όλε αυτέ τι τις ad hoc προσπάθειε και θα πρέπει να περάσει ο χειρισμό εξόδου ξεκαθαρίσει το τοπίο. Τώρα για την Σρι Λάγκα. Έχω συντάξει εγώ και η Καφιάστον μία επιστολή και λέμε ότι μελετούμε τη δυνατότητα παρέκτασης και παράτασης της σχετικής περίοδου. Αναστολή ακόμα ένα εξάμεινο. Πώς είναι αυτά τα benchmark, αυτά τα κριτήρια. 12. Τον Ιούλιο. Είπαμε θα το αποφασίσουμε. Να, μια δεύτερη ευκαιρία που τους δίνουμε. Με αυτά όλα τα benchmarks. Όλα αυτά ξεκάθαρα και τον Ιούλιο θα κρυφτεί το θέμα. Με ευρύτατες διαβουλεύσεις. Με την κυβέρνηση της χώρας κλπ. Άλλη ερώτηση. Κύριο Ντίβα από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Δεν ξέρω πως πρέπει να έχουμε ε, ανώνυμες παρατηρήσεις γιατί θα πει ο κόσμος περισσότερα. Δεν είναι, έχω αντίρρηση με αυτό. Να μπορεί ο κόσμος αν θέλει μόνο να δημοσιεύει το όνομά του. Δεν έχω καταλήξει. Θα το κοιτάξω και θα σας πω. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ και θα ήθελα 4,5 να κλείσουμε. Όμως, ακόμα, διάφοροι έχουν ζητήσει το λόγο. Πέντε και παραπάνω, οπότε θα πρέπει να μπει ένα χρονικό όριο. Πρώτη η Κριστιάνα Μουσκαρντίνη του ΕΛΚ. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Επιτροπό του για την απάντηση για τη Σρι Λάνκα. Να θυμηθήσω, ωστόσο, ότι η Σρι Λάνκα είχε προεδρικές εκλογές τον Γενάρη και κοινοβουλευτικέ την Άνοιξη. Είναι δύσκολο, λοιπόν, μέχρι την 1η Ιουλίου να έχουν φτάσει σε θέση να αλλάξουν την ε, πορεία τους και την κατάσταση της χώρας που από χρόνια είναι πολύ δυσχερής. Η δική μα λοιπόν πρόθεση είναι να ζητήσουμε από την Επιτροπή να παρατείνει ω το τέλο τη χρονιά την αναστολή, ώστε αυτή η χώρα να μπορέσει να φτάσει στο επίπεδο που πρέπει. Έπειτα, ο επίτροπο σωστά ανέφερε για το, άνοιγμα νέων αγορών. Για να διερευνήσουμε και να ανοίξουμε όμω νέε αγορέ, κύριε Επίτροπε, πιστεύω θα πρέπει να έχουμε υπόψη και αυτό που το Ευρωκοινοβούλιο έχει εκφράσει από την προηγούμενη ήδη θητεία για την διεθνοποίηση δηλαδή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο να ανοίξουν οι αγορέ εάν οι δικέ μα μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει τη Ευρώπη δεν έχουν δυνατότητα πρόσβαση σε αυτέ τι αγορέ. Το εξετάσουμε δηλαδή, όπω έκανε και το Κοινοβούλιο, τα διάφορα προσκόμματα για την ε, έξοδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ευρώπης στις υπόλοιπες αγορές είναι σημαντικό. Και σε ό,τι αφορά τώρα την οικονομική βιωσιμότητα, αυτή η βιωσιμότητα θα πρέπει να οδεύει παράλληλα με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Ιδάλλως, απειλούμεθα να έχουμε μια εικονική βελτίωση της κατάστασή μας και σε μερικά χρόνια να, να αντιμετωπίσουμε σοβαρότατα πλήγματα. Να θυμίσω μόνο αυτό που συνέβη στην Αφρική. Έτσι ως παράδειγμα. Και να αναφέρω εδώ και το πρόβλημα του πακέτου που αναφέρεται για τα τελωνία και τον εναρμονισμό. Πρέπει να φροντίσουμε να γίνει αυτό σύντομο, ώστε να ρεποδίσουμε και την εισαγωγή παράνομων εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ερώτησή μου αφορά τη σχέση και τη συνεργασία της εξωτερικής πολιτικής με το εμπόριο. Έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα και μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση υπόψη. Βάσει της πρόσφατης νεοθεσπιστής σας διαδικασίας θα πρέπει το Κοινοβούλιο να δίνει την συγκατάθεσή του για τη συμφωνία σύνδεσης με οποιαδήποτε χώρα και συγκεκριμένα με το Ισραήλ. Αυτήν την εβδομάδα άκουσα κάποιες ομάδες στο Ευρωκοινοβούλιο θέλουν να παγώσουν την έγκριση της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών με το Ισραήλ. Εδώ βεβαίως υπάρχει κάποια, είναι αμφιλεγόμενο το ζήτημα ακριβώ λόγω των απολειών ε, ζώων στις, ε, στη Λόρδα της Γάζας και λόγω των δράση των ένοπλων δυνάμεων του Ισραήλ. Πιστεύετε κύριε Επίτροπο ότι θα πρέπει αυτή η συμφωνία να παγώσει ή να αναβληθεί για πολιτικούς λόγους και επίση, ποιε θα ήταν ενδεχομένω οι επιπτώσει. Και τέλο, θα μπορούσαν το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσουν σε ισχύ την συμφωνία στο και προσωρινά, εάν τυχόν διαφωνήσει το Κοινοβούλιο. Είναι, επαναλαμβάνω, δυνατό το Συμβούλιο και η Επιτροπή να προβλέψουν προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας. Εάν το Κοινοβούλιο θελήσει να παγώσει την έγκριση, να αναβάλει δηλαδή την έγκρισή της. Να ευχαριστούμε ο κύριος Χέλιν από το ΕΛΚ. Κύριε Επίτροπε, η εμπορική πολιτική είναι διάσημη για πάρα πολλά. Όμως εδώ έχουμε υπόψη την πρωτοβουλία τα πάντα εκτό από όπλα. Everything but arms. Θα σα παρακαλούσα λοιπόν το μέλλον τη εμπορική πολιτική να μην γίνει στο μέλλον everything but trade, τα πάντα εκτό από εμπόριο. Μα με βάση αυτά που μας είπατε σήμερα, ε, είδαμε ότι δεν είναι έτσι, αλλά μη γίνει η εμπορική πολιτική ομπρέλα και όλες τις άλλες πολιτικές. Μην γίνει δηλαδή ένα μέσο για να καλύπτουμε όλα τα άλλα εκτός από το εμπόριο τελικά. Και στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020, να πω για τις ασφαλείς ευρωπαϊκές επενδύσεις στο εξωτερικό. Ε, το πλαίσιο για τις μελλοντικέ μας συμφωνίες πιστεύω είναι καθοριστικό. Εδώ η ανησυχία μου είναι, αν και δεν έχουμε δει ακόμα την πρόταση, πού θα επικεντρωθεί η Επιτροπή. Δηλαδή, να ε, πάυσουν οι διμερεί επενδυτικέ συμφωνίε των επιμέρους κρατών μελών. Καταλαβαίνω ποιοι είναι οι λόγοι που μπορεί εδώ να υποκρύπτονται, αλλά νομίζω πιο σημαντικό είναι να ε, καθορίσουμε ένα πλαίσιο για μια ισχυρή ανταγωνιστική ευρωπαϊκή επενδυτική πολιτική. Όχι να κοιτάξουμε πώς θα πάυσουν, θα τερματιστούν οι διμερείς συμφωνίες των κρατών μελών. Είναι σημαντικό να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική και σε συνεργασία με τι κυβερνήσει των χωρών και με τα θεσμικά όργανα. Γιατί οι εταιρείε τη Ευρώπη χρειάζονται ασφάλεια. Μπορείτε να μα δώσετε λοιπόν κάποιε ιδέε, σχόλια σε αυτό το τομέα. Εδώ αυτό πραγματικά με απασχολεί ιδιαίτερω. Ευχαριστούμε κύριο Χίγκιν από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, να σας ρωτήσω τι αλλαγές προβλέπετε στην εμπορική πολιτική και στη στρατηγική της σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης της χιλιετίας, η εκρίζωση της ακραίας φτώχειας και πείνας και η μείωση της παιδικής συνεισιμότητας είναι μόνο δύο παραδείγματα και αυτά είναι άμεσα συνδεδεμένα με την εμπορική διάσταση. Ποια είναι τα δικά σας προγνωστικά. Τι θα γίνει με τον κίνδυνο μιας νέας ε, ύφεσης. Τι προβλέπετε εσείς και το ευρύτερο θέμα της σχέσης του εμπορίου με τις δραστηριότητες ε, των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Μπαρόζο και τη Επιτροπής στην οποία εσεί ανήκετε, είναι σαν να έχουν δράσει υπέρ των κερδοσκόπων στις χρηματοπιστωτικές αγορές τους. επιτρέψατε να εκβιάσουν τις οικονομίες χωρών όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Και η Επιτροπή απαιτεί οι μισθοί των εργαζομένων και τα ωφελήματά τους να περικοπούν ακριβώς εξαιτίας των, ετοιμάτων των αιτημάτων των χρηματοπροστατικών ε, αγορών. Τα δισεκατομμύρια λοιπόν που αποστραγγίζουν από τις εθνικές οικονομίες αυτά τα παράσιτα είναι δισεκατομμύρια τα οποία δεν θα τα, τα, τα ξοδέψουν τελικά αυτοί οι άνθρωποι σε υπηρεσίες και προϊόντα. Άρα δεν θα προωθηθεί το εμπόριο. Βλέπετε λοιπόν εδώ την αντίφαση. Και το ερώτημά μου είναι συγκεκριμένα γιατί πιέζεται τόσο την Αμήμπια ώστε να υπογράψει ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής συνεργασίας προτού η Αναπτυξιακή Επιτροπή του Κοινοβουλίου της Νοτιού Αφρικής διαβουλευτεί μαζί μας. Γιατί γίνεται αυτό τώρα. Έχετε λάβει πολλές επιστολές από μη κυβερνητικέ οργανώσεις για το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ε, καλημέρα σας, δεν σας έχω χαιρετήσει ακόμη. Καταρχήν ε, χαίρομαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά μία διαβούλευση για την ε, εξωτερική εμπορική πολιτική η οποία θα ολοκληρωθεί στις 28 Ιουνίου και όλες οι χώρες και όλα τα άτομα μπορούν να απαντήσουν στα ερωτήματα αυτά και να εμπλουτίσουν τη συζήτηση. Αλλά τα θέματα αυτά και τα έγγραφα τα οποία προτείνονται θα έπρεπε πέραν των αγγλικών να είναι και σε άλλες γλώσσες να μπορούν να απαντήσει περισσότερος κόσμος. Επίσης ε, μιλάμε για την ε, συνοχή της ε, μορικής πολιτικής με την κοινωνική, την γεωργική και ούτω καθεξής. Αλλά ξεχνάμε συχνά τη σχέση μεταξύ της μορικής πολιτικής και της έρευνας. Ορισμένοι θεωρούν ότι υπάρχουν ανοιχτές αγορές και μπορούν να πουλήσουμε ε, προϊόντα εφόσον υπάρχει μεταφορά τεχνολογική, τεχνολογικών γνώσεων. Αλλά βλέπουμε ότι ε, το κενό το οποίο ενδεχομένως υπήρχε στο παρελθόν ε, μειώνεται και πάει. Μήπως λοιπόν εσείς σαν Επίτροπος Εμπορίου και άλλοι επίτροποι σκέφτεστε τι θα γίνει εφόσον πλέον δεν θέλει η Ευρώπη να επενδύει τόσο στην πολιτική έρευνα ε, Τα άλλα θέματα περί περιβάλλοντος ε, τα αναφέρατε προηγουμένως. Είπατε να μην είμαστε πολύ σκληροί και να υπάρχει περισσότερη ευελιξία. Αλλά θα μπορούσαμε συγχρόνως να είμαστε προοδευτικοί σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ε, κοινωνικές επιταγές. Βλέπουμε δε ότι το άτομο εξαφανίζεται στην εμπορική πολιτική ε, από τα κράτη. Ε, μήπως λοιπόν θα μπορούσαν στο μέλλον τα μεμονωμένα κράτη να έχουν περισσότερη εμπλοκή στα θέματα αυτά και όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον είστε ο αρμόδιος επίτροπος. Καταρχήν ήταν η, κυρία, η ερώτηση της κυρίας Αντρικιένε. ή στις ε, συμφωνίες δεν προβλέπεται ε, εφαρμογή. Σε ορισμένες παραδείγματος χάρη ε, προβλέπεται μία τέτοια ρήτρα, όχι σε άλλες. Αν είναι κάτι παγωμένο, είναι παγωμένο και δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα από αυτού. Ο κύριος Φέλνερ είπε προκλητικά ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο το εμπόριο αλλά υπάρχουν και άλλα δικαιώματα ε, κοινωνικά και άλλα. Ότι πέραν ε, του, εμπορικού, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που γκρινιάζει και το Συμβούλιο γκρινιάζει διότι βλέπουν ε, ότι παραδείγματος χάρη όσον αφορά τις σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες για να φέρω ένα παράδειγμα βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο προφανή. Όσον αφορά τις επενδύσεις Υπό μαλά συνθήκα στην επόμενη εβδομάδα η ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα υιοθετηθεί από το Κολέγιο των ε, Επιτρόπων. Είναι ένα θέμα που συζητείται. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές διαφωνίες, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση. Θα δείτε λοιπόν την ανακοίνωση την άλλη εβδομάδα σε τρία τμήματα και Υπάρχει και ένα σύστημα εξουσιοδοτήσεων που τα κράτη-μέρη μπορούν να διαπραγματευτούν μεμονωμένα και ε, υπάρχει και ένα προοδευτικό κομμάτι. Αλλά θα χρειαστεί να βρούμε τέρους για να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό και εξαρτάται και από τα κράτη-μέλη. Και έτσι έρχομαι στο τελευταίο ερώτημα του κυρίου Αρίφ για τα ε, κοινοτικά συμφέροντα σε σχέση με αυτά των κρατών μελών. Μπορούμε να προχωρήσουμε εάν τα κράτη-μέλη συμφωνήσουν ότι πλέον δεν θα βασίζονται στις μεμονωμένες συμφωνίες αλλά θα υπάρξει μία κοινή στρατηγική. Είναι μία πολιτική συζήτηση την οποία προωθούμε πολύ σκληρά. Όσον αφορά τη Σρι Λάγκα, κυρία Μουσκαρδίνη, σας είπα τι θα κάνουμε, de facto, εάν υπάρξει μία αποδεκτή απάντηση πριν της 1ης Ιουλίου θα υπάρξει μία επέκταση μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Αλλά πρέπει να αντιδράσουν. Αν δεν αντιδράσουν τότε θα χρειαστεί να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και προς την άλλη κατεύθυνση. Υπάρχουν δηλαδή πολλά τα οποία μπορούν να γίνουν. Όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την πρόσβαση στις αγορές, ε, είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε γιατί είναι κρίσιμο για την ευρωπαϊκή οικονομία. 90% των ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες και μπορούμε να μάθουμε πολλά και να διδαχθούμε από την έκθεση που έχει καταρτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά την οργάνωση των τελωνίων δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα την ερώτηση αυτή γιατί νόμιζα ότι υπάρχει μια τελωνιακή ένωση. Ενδέχεται όμως να υπάρχουν διαφορές και είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να θέσετε στον αρμόδιο υπουργό τον κύριο Σεμέτα. Κύριε Χίγγινς, δεν είναι πρώτη φορά που καταλήγω στο συμπέρασμα ότι έχουμε ουσιαστικές διαφορές απόψεων μεταξύ μας μεταξύ πολιτικής ε, και ε, ε, εμπορικής πολιτικής αλλά και αυτά είναι μέρη της της δημοκρατικής διαδικασίας. Δεν μπορώ να σας πω ότι εγώ διαφωνώ με όλες τις απόψεις σας. Ενδεχομένως όμως εσείς μου είπατε γιατί δεν πιέσαμε την Ναμίμπια να υπογράψει πιο νωρίς. Δεν είναι θέμα της Ναμίμπια, αλλά υπάρχουν τρελές καταστάσεις στην ε, ε, Αφρική όπου έχουν μονογραφηθεί ορισμένες συμφωνίες και μετά δεν υπογράφονται και αναρωτιέται κανείς ε, αν υπάρχει νομική βάση για να συνεχίσει να προωθείται μία προτιμησιακή σχέση και νομικά το ερώτημα είναι πολύ ορθό. Δηλαδή δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο περιερίζεται στην Αμίμπια αλλά και σε πολλές άλλες χώρες ε, της Αφρικής και θα χρειαστούν ίσως μήνες πολύ για να καταλήξουμε σε μία λύση. Η μεταφορά. Ε, ε, εάν ε, πρέπει να επεκταθούμε στην έρευνα διότι διαφορετικά θα περιοριστεί η τεχνολογική μας πρόοδος. Όντως το συζητάμε ιδίως σε σχέση με την Κίνα. Εύχομαι διότι οι προτάσει σαν την Indigenous ε, Innovation, ε, ε, υποχρεωτική πιστοποίηση και με ανησυχεί πάρα πολύ το καθεστώς. Όχι τόσο η δημοσίευση των, των γνώσεων, αλλά η η Κίνα θα προχωρήσει τόσο πολύ ε, στα επόμενα χρόνια που θα πρέπει να έχουμε μόνοι μας δυνατότητες ε, επαρκής. Ε, υπάρχουν τόσα πολλά ερευνητικά εργαστήρια στην Κίνα που αναρωτιέται κανείς αν θα μπορούμε στο μέλλον να εξάγουμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας και η εμπορική πολιτική της Κίνας είναι κάτι το οποίο θα αξίσει να συζητηθεί στην Επιτροπή αυτή. Αλλά από όλους τους φακέλους τους οποίους ε, ε, έχω αναλάβει αυτός με ανησυχεί περισσότερο από όλους. Ευχαριστώ. Φτάσαμε στο τέλος της ε, συζητήσεώς μας. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε και μας Παρουσιάστε τις ιδέες σας για την επόμενη ε, ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική του 2020. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε λιγότερο από ε, δύο ώρες και πρέπει να επεξεργαστούμε ε, πέντε ακόμη θέματα, άρα λιγότερο από μισή ώρα το καθένα. Λοιπόν, χωρίς να καθυστερούμε, ας προχωρήσουμε στο σημείο 12. το 12 η θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού όπως το έχει τροποποιήσει το Συμβούλιο. Είναι μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ο υπεύθυνο εισηγητής είναι ο Πίτερ Στάσνη του ΕΛΚ και αποφασίστηκε να γνωμοδοτήσουμε προς την Επιτροπή Προπολογισμού. Πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι εδώ ο εισηγητής. Οπότε θα ζητήσω από τον Ντάνιελ Γκάσπαρη να παρουσιάσει το θέμα αυτό για αυτόν. Ε, αξιότιμε ε, κύριε ε, Πρόεδρε, ο, ο, με παρακάλεσε να παρουσιάσω τα, το θέμα αυτό και βλέπουμε ότι υπάρχει μία πρόταση για 142 δισεκατομμύρια σε μία αύξηση σε σχέση με το 2007 και ε, σε άλλα θέματα μία αύξηση στάξεως ε, ε, του 5,5% υπάρχουν γενικές ε, ε, δεσμεύσεις ε, ιδίως για την γεωργία και άλλες για πληρωμές και ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά 64,4 δισεκατομμύρια θα αφιερωθούν για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πράγμα το οποίο θα είναι ευπρόσδεκτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία επλήγει από την δημοσιοοικονομική ε, κρίση. Υπάρχει μία γενική αύξηση 12,8% και οι πληρωμές επίσης αυξάνονται κατά 15%. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ότι 12,6 δισεκατομμύρια ε, δεσμεύσεων έχουν περιληφθεί και η πρόταση για το 2011 είναι 250 εκατομμύρια ευρώ διότι ε, υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες ε, ε, ζητούν βοήθεια και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει η τάση αυτή και τα επόμενα έτη. Ξέρετε ότι η πρόταση για το ICI δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί και μιλάμε επιπλέον για 25 δισεκατομμύρια ευρώ ε, για να προωθηθεί το πρόγραμμα TCI και τέλος ε, θα υπάρξει μία αύξηση ε, και των οικονομικών προγραμμάτων. Επίσης ε, θα χρηματοδοτήσουμε ένα πρόγραμμα στην Ινδία, ένα στην Ταϊλάνδη, ε, θα εξυπηρετήσουμε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις το ταχύτερο δυνατόν και προσωπικά θα ήμουν πολύ ευτυχής αν κάποια μέρα μπορούσαμε να μιλήσουμε και στη δικιά μας Επιτροπή για αυτά τα ευρωπαϊκά επιχειρησιακά κέντρα. Όσον αφορά το Κοινοβούλιο, νομίζω ότι είναι προφανές ότι έχουμε δυνατότητα δυνατότητα να συμβάλλουμε στην πολυμερή συνεργασία στα πλαίσια του ΠΟΕ, ιδίως μέσω της διασκέψεως και των ομάδων εφόσον υπάρχουν οι πόροι και πρέπει να τονίσουμε ότι η Επιτροπή Ίντα έχει μπει σε μια καινούργια φάση στη συνέχεια της Συμφωνίας της Λισαβόνας και γι' αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι πόροι θα διατίθενται για να ανταποκριθούν εις ε, τις ε, ανάγκες της Επιτροπής μας που γίνεται όλο και πιο σημαντική. Αυτά είχα να σας διαβάσω εν ονόματι του εισηγητή Πίτερ Στάζη και μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση. Ο δε Πίτερ Στάζη ευχαρίστως θα συνεργαστεί στενότατα με τους συναδέλφους εάν του το ζητήσουν. Θέλετε να συζητήσουμε το θέμα αυτό, Ευχαριστούμε τον Ρόμπερ και το έργο που έχει κάνει και ελπίζουμε να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια αποτελεσματικά. Απλώ να επιστήσω την προσοχή σα σε δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα το Ταμείο Παρακολούθηση τη Αγορά τη Μπανάνα. Σήμερα υπάρχει και συζήτηση για το θέμα τη μπανάνα. Θα πρέπει να αποφανθούμε σύντομα για τη σύναψη συμφωνία στον ΠΟΕ για το εμπόριο μπανάνα η συμφωνία αυτή μπορεί να ικανοποιεί τι χώρε τη Λατινική Αμερική και τι χώρε τη Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν θα περάσω τώρα στι λεπτομέρειε του, του όλου θέματο και τι ανάγκε τη χώρα των χωρών ΑΚΕ. Όμω εδώ με τα συνοδευτικά μέτρα που έχει προτείνει η Επιτροπή υπάρχει ένα διπλο, διτό πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα το χαρτοφυλάκιο είναι πολύ χαμηλό, 100 εκατομμύρια ευρώ για τρία χρόνια για όλε τι χώρε ΑΚΕ δεδομένου ότι οι εξαγωγέ μπανάνα για ορισμένε χώρε είναι μόνη πηγή εισοδήματο και απασχόληση, για την Γουαδελούπη λόγου χάρη, και έπειτα το, τα κονδύλια που θα χρηματοδοτήσουν το πρόγραμμα αυτό θα προέρθουν από αναπτυξιακά προγράμματα που απευθύνονται αρχικά σε άλλους τομείς. Ο κινησμό τη επιτροπή να πάρει τα κονδύλια αυτά και να χρηματοδοτήσει την αγορά τη μπανάνα από άλλα προγράμματα, όπω τη καταπολέμηση των ασθενών που προέρχονται από τη φτώχεια, ε, αυτά όλα μα θέτουν ε, ερωτήματα δεντολογικά. Πρέπει εδώ να γίνει κάποιο ξεκαθάρισμα και νομίζω ότι χρειάζεται να γίνει συζήτηση για τη χρηματοδότηση αυτή και έπειτα για τι εμπορικέ βοήθειε. Εδώ και χρόνια ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι εμπορικέ επιδοτήσει συγκεκριμένου αριθμού και παίρνουμε μόνο μερικέ απαντήσει, καμία συγκεκριμένη. Θέλουμε ανά χώρα να ξέρουμε τι γίνεται με τις εμπορικές επιδοτήσεις. Για τα δύο αυτά σημεία λοιπόν, τουλάχιστον ως προ τον προπολογισμό, θα πρέπει να έχουμε κάποιες διευκρινήσεις. Και ελπίζω ότι στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων θα έχουμε την ευκαιρία να θίξουμε και άλλα θέματα. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχετε να απαντήσετε κάτι στα ερωτήματα που τέθηκαν η κυρία Σεσίλ Μπιλό. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή που δεν είναι ο ίδιος εδώ, αλλά θα αναλάβει τη σύνταξη της έκθεσης και τους βουλευτές που έκαναν τα σχόλιά τους. Στην πρώτη μου αυτή σύντομη παρέμβαση θέλω να τονίσω ότι σε ό,τι αφορά την συνέχεια του προπολογισμού για τα εμπορικά θέματα τα τελευταία χρόνια, βεβαίω θα επικεντρωθούμε στην ανάκαμψη στον ευρωπαϊκό προπολογισμό μα, όπω σωστά επεσήμανε ο εκπρόσωπο του εισηγητή. Οι περισσότερε αυξήσει εντοπίζονται στο κεφάλαιο 1 και 2. Τώρα για το συγκεκριμένο ερώτημα για το Ταμείο τη Μπανάνα, Ακόμη μιλάμε για το σχέδιο προπολογισμού του 2011 και είναι αποτέλεσμα της συμφωνίας που συνήθισε στα τέλη του 2009. Οπότε η χρηματοδότηση έχει οριστεί με βάση αυτή τη συμφωνία. Για το άλλο σας ερώτημα, σε ό,τι αφορά την βοήθεια για το εμπόριο, Aid for Trade, υπάρχει ετήσια έκθεση που ετοιμάζει η Κομισιόν ούτως ή άλλως για, για το Aid for Trade και για το πώς δαπανώνται τα κονδύλια αυτά. Μιλάμε για ένα στόχο των 2 δις βάσει της επίσημης έκθεσης που νομίζω δημοσιεύτηκε πριν από δίμηνο. Στόχος λοιπόν των δύο δις επετέχθη και η αύξηση στις δαπάνες του προγράμματος Aid for Trade αφορά κυρίως τις χώρες ΑΚΕ αύξηση τάξη του 36%. Βεβαίω είναι δύσκολο να έχει κάνει ε, όλε τι λεπτομέρειε όλου του προγράμματο, γιατί το Aid for Trade, ε, η βοήθεια για το εμπόριο, είναι μέρο τη συνολική μα αναπτυξιακή πολιτική και των ανάλογων ε, σχέδιων τη Επιτροπή. Πάντω σημειώνουμε τα σχόλιά σα και θα φροντίσουμε να επανέλθουμε στο θέμα αυτό στο πλαίσιο της συνέχεια της ανταλλαγής απόψεων που θα γίνουν εδώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κάποια συμπεράσματα από τον κύριο Κάσπαρη εκ μέρους του εισηγητή. Ωραία λοιπόν, θα αναμένουμε το σχέδιο γνωμοδότησης σε μια ύστερη χρονική στιγμή. Περνάμε τώρα στο σημείο 13. Ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Η εισηγήτριά μα είναι η κυρία Τοκία Σαΐφη από το ΕΛΚ και θα της δώσω το λόγο. Χωρίς να κάνω προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν ξεκινήσω, να διευκρινίσω ότι το χρονοδιάγραμμα έγκριση αυτή τη έκθεση είναι συμβατό με το χρονοδιάγραμμα του, του προγράμματο κ. Ντεζίρ για τις κοινωνικέ ευθύνες των επιχειρήσεων και επειδή τα δύο θέματα αυτά μπορούν να εξεταστούν συγχρόνω, είναι αλληλένδετα. Να ευχαριστήσω μάλιστα τον κύριο Ντεζίρ που δεν είναι παρόν για τη συνεργασία, για τη συνεργασία του. Να, δεν θα σα κάνω σήμερα μια συνολική παρουσίαση του θέματο, διεξοδική, αλλά ήθελα να θίξω την πολιτική διάσταση τη συμφωνίας αυτή. Όπω ξέρουμε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εφαρμογή των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων στι διεθνεί εμπορικέ διαπραγματεύσει, είναι ένα θέμα πολύπλοκο. Από τη μια οι χώρες του Βορρά καταγγέλουν το περιβαλλοντικό και κοινωνικό ντάμπινγκ κάποιων αναδυόμενων χωρών. Από την άλλη οι χώρες του Νότου υποψιάζονται τις χώρες του Βορρά ότι έχουν παρεμποδίσει την οικονομική τους ανάπτυξη και με την απέτηση να υλοποιούνται αυτές οι ε, προδιαγραφές ασκούν ένα μέρος ε, ύπουλου προστατευτισμού και καλυμμένου προστατευτισμού. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε τι θέλουμε για την εμπορική πολιτική του αύριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενία, τα εννέα πρότυπα σε θέματα ασφάλειας, ε, υγείας, και προστασία των εργαζομένων των καταναλωτών, καθώ και του περιβάλλοντο, μα δίνουν ένα συγκεκριμένο ευρωπαϊκό μοντέλο, ένα ευρωπαϊκό πρότυπο, το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ω πηγή έμπνευση σε διεθνέ επίπεδο και στι πολυμερεί μα διαπραγματεύσει. Η δική μας επιθυμία σήμερα είναι να δούμε θετικά την όλη έκθεση. Δηλαδή, να καταλάβουμε ότι από τη μια πρέπει να γίνονται σεβαστές οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές και Επίσης, ε, οι εμπορικές ανάγκες, ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία να συμβάλλουμε σε μια επανειδιοποίηση, θετική μάλιστα, της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία θα μπορούσαν να εκλάβουν διαφορετικά οι πολίτες και να ενισχύσουμε την ε, συζήτηση για την ανταλλαγή απόψεων. Η συμφωνία αυτή θα αποτελείται από, τρεις, από τρία βασικά κεφάλαια, τα πολυμερή, τα μονομερή και τα διμερή. Κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα κάποιες ιδέες για να οργανώσουμε τη συζήτησή μας. Στο πλαίσιο το πολυμερές η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να περασπιστεί την πρόθεση της αξιοπρεπούς εργασίας και να παροτρύνει τους συνεργάτες της να υπογράψουν και να κυρώσουν τις οκτώ συμβάσεις, τις βασικές συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας. Επίσης θα πρέπει ένας οργανισμός όπως το Παγκόσμιο, Οργανισμό, το Οργανισμός Εργασίας έχει ένα μια υπηρεσία έγκριση των προδιαγραφών και να φροντίζει την ε, επιβολή τους για τις νομικές και κοινωνικές ε, προδιαγραφές. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια δυνατότητα εξέταση προδικαστικών ερωτημάτων από τον ΠΟΕ και να εξετάζονται από το Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασία και αυτό λόγω χάρη για κάποιε από τι πρημοδοτήσει. Τώρα, στι διμερεί συμφωνίε θα πρέπει να σκεφτόμαστε την ε, υποκείμενη σε προποθέσει απελευθέρωση, όπως λόγου χάρη την ε, σταδιακή άρση των φραγμών ή την υποπροποθέσεις πρόσβαση στην αγορά, αναλόγως με το σεβασμό και την τήρηση της μια τη άλλη υποχρέωση για ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικέ και περιβαλλοντικές ε, προδιαγραφές. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει και η διακύμανση, η δυνατότητα μεταλλαγή της αποτίμησης της κατάστασης των διαφόρων χωρών ανάλογα με το πώς γίνονται σεβαστές οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές ρήτρες καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και επίσης στο πολυμερές επίπεδο στην μεταρρύθμιση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων θα πρέπει να σκεφτούμε εδώ τους δικαιούχους λαμβάνοντας υπόψη το αναπτυξιακό τους επίπεδο και διασφαλίζοντας μια πλήρη παρακολούθηση του κατά πόσο ανεπληρώνουν τις δεσμεύσεις σε αυτόν τον τομέα. Σε γενικές γραμμές προτού έχουμε γενικές ε, διαθέσεις και έγκριση φιλόδοξων σχεδίων θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια μετρημένη εδώ πολιτική επιτρέποντας να θεσπίσουμε ένα σύστημα διεθνούς εμπορίου δικαιότερο. Ιδού, Πρόεδρε, εντάχει οι πρώτες μου παρατηρήσεις. Θα είμαι βεβαίω στη διάθεση των συναδέλφων για να ακούσω και τα δικά του σχόλια. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. Ανοίγουμε τη συζήτηση και δίνω το λόγο στον David Μάρτιν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια και ελπίζω ότι τελικά θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια συνένεση οι πολιτικές ομάδες στην Επιτροπή μας. Πρώτα-πρώτα θέλω να σας πω ότι όποτε μιλάμε για Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου κάνουμε την μελέτη των οικονομικών επιπτώσεων. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να γίνεται και μια αποτίμηση των επιπτώσεων στα ανθρωπίνα δικαιώματα ούτως ώστε να ξέρουμε ποια είναι τα πραγματικά αποτελέσματα μιας ε, τέτοιας συμφωνίας. Να, για παράδειγμα, πάρτε την Κολομβία. Ίσως έχει δίκιο η Κομισιόν, δεν ξέρω, που λέει ότι εάν διαπραγματευτούμε με την Κολομβία, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Άλλοι μας λένε όμως ότι έτσι αμείβουμε μια κακή επίδοση των ανθρωπίνων δικαιώματων. Εγώ σας λέω ότι θα πρέπει κάποιος ε, αμερόληπτος να κάτσει και να ζυγίσει τι ισχύει, τι επιπτώσεις θα υπάρχουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα όσον αφορά τα περιβαλλοντικά πρότυπα, το κάνουμε αυτό με την Κορέα, θα πρέπει όμως να δούμε τι γίνεται με την κοινωνία των πολιτών, Ιδίω αφού δίνουμε σε κάποιον τα μέσα να οργανωθεί όπως την κοινωνία των πολιτών. Μια που κάτι τέτοιο πρώτα πρώτα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα για το σύστημα γεννημένων προτιμήσεων, πλάς, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι κανείς έχει αυτό το στάτους εάν προσυπογράψει τα κείμενα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ή Αυτό σημαίνει όχι μόνο ότι μένει τιμόρυτος κάποιος ο οποίος δεν θα τηρεί τις υποχρεώσεις του, αλλά σημαίνει και το ότι κάποιος άλλος που κάνει το σωστό δεν αμείβεται και αδικείται. Άρα θα πρέπει να υπάρχει σωστή επιτήρηση και εποπτεία επίσης. Αυτά έχουν ζητήσει βέβαια και σε άλλες επιτροπές του Κοινοβούλιο για τα βασανιστήρια και όπως για το θέμα των ευρωπαϊκών εταιριών που δίνουν υλικό για μπλοκάρισμα του διαδικτύου και συναφή φαινόμενα που έχουν γίνει κατά συρροή θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και ποιες χώρες χωρίς να το ξέρουν δίνουν τέτοια όργανα μέσα καταστολής δημοκρατικών ε, δραστηριοτήτων σε κάποιες τρίτες χώρες. Uh, Τέλος για τους πρασίνους. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αυτή είναι η πρώτη μου παρέμβαση εδώ στην ε, Επιτροπή. Ελπίζω να μπορέσω να σας βοηθήσω, είναι θετική συμβολή μου και θα ήθελα πρώτα-πρώτα τη, γνώση, τη, τη, τη, γνώμη και άλλων επιτροπών ε, για να μας πούνε τη γνώμη τους αυτές οι επιτροπές των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των περιβάλλων πώς τα βλέπουν τα εμπορικά πώς γίνεται δηλαδή να έχουμε κάποιον ε, κώδικα διοντολογίας που χωρίς να είναι υποχρεωτικός να είναι αποδοτικός δεν γίνεται αυτό ήδη πράσινη θα θέλαμε να υπάρξουν κάποια μέτρα πρώτα πρώτα τα κεφάλαια, τα σχετικά με την αηφορία στις συμφωνίες εμπορικές θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά, θα πρέπει να υπάρχουν στη δικασία λύση ε, διαφορών επίσης η μελέτε των επιπτώσεων. Πολλέ φορέ ολοκληρώνονται πριν κλειστεί η συμφωνία. Όμω, πολλέ φορέ αυτά τα οποία περιέχουν σαν συμπεράσματα δεν οδηγούν στην ε, συμπερίληψή του στι τριγωνικέ συνθήκε. Άρα, θα πρέπει για να είμαστε εντάξει να εξασφαλίσουμε ότι οι διαπραγματεύσει ακολουθούν αυτές τις επιπτώσεις. Επίσης η αξιολόγηση των ε, επιπτώσεων των αυτών των ε, συμφωνιών για τους εργαζόμενους και το περιβάλλον θα πρέπει να γίνονται σε συνεργασία με συνδικαλιστές, με μη κοινωνικούς οργανισμούς. Επίσης οι εμπειρογνώμονες και αυτοί θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να βοηθούν στην διόρθωση των τυχών λαθών. Τέλος, οι προτάσεις του του ειδικού εκπροσώπου του ΟΗΕ για ανθρώπινα δικαιώματα και επιχειρήσεις protect, respect και remedy θα πρέπει αυτά προστασία, σεβασμός και επανόρθωση όλα αυτά θα πρέπει να ενταχθούν στην πολιτική μας επίσης θα πρέπει νομίζω η Κομισιόν να μας διαφορήσει όσον αφορά τα εξής η Σουηδική Ισπανική Προεδρία είχαν εισαγάγει τον του 2009 κάποιες ρήτρες στις διαπραγματεύσεις. Για κάποιες προσωρινές συμφωνίες, ε, τι έγινε από τότε, τι έγινε με, με, με αυτές τις δεσμεύσεις, το CSR. Θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται. Πώς θα μπορέσουμε και αυτές τις συμφωνίες, δεν μπορούμε να τις υπαγάγουμε στους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών. Συνήθως αγώνας λέει ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ρυθμίσει τα των επενδύσεων. Θα πρέπει αυτό να καλύπτει στο σχετικό κανονισμό της Κομισιόν να καλύπτει και τις υποχρεώσεις των επενδυτών. Και περιμένω πώς και πώς τη συνέχεια της εργασίας της συγκήτριας. Ευχαριστούμε και καλώς στην Επιτροπή μας, λέει ο Πρόεδρος. Ελπίζω ότι αυτό πρόκειται να σας ε, βοηθήσει. Τώρα, παρακολουθήστε το χρονικό όριο. Ευχαριστώ πρώτα. θα είμαι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Πολλές φορές οι βουλευτές είμαστε αφελείς, αισιόδοξοι. Και αυτό αφορά και τους κανόνες ε, δικαίου για περιβάλλον και κοινωνική πολιτική. Τα άκουσα αυτά στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων, αλλά παρόλα αυτά φοβάμαι ότι τα ίδια λέμε συνέχεια. Ενώ έχει παιχτεί το παιχνίδι. Να σας εξηγήσω. Έχω την εντύπωση ότι η Κομισιόν λέει ότι θέλει το Κοινοβούλιο να βάλουμε ένα σωρό πράγματα να βάζουμε στις συμφωνίες εμπορικές και πρόκειται να τους ικανοποιήσουμε τους ε, Ευρωβουλευτές. με άλλη μεριά είναι οι χώρες του Νότου που έχουν την ίδια λογική και λένε οι Ευρωπαίοι πρέπει να καθησυχαστούν όσον αφορά τι ε, διεθνείς συμφωνίες ε, υπό τον όρο προστασίας των δικαιωμάτων και τήρησής τους. Από την άλλη μεριά όμως, ούτε αυτές οι χώρες, ούτε η Κομισιόν όμως α, υποχρεούνται να τηρήσουν τα υπεσχημένα. Γι' αυτό και σας λέω ότι όλη αυτή η κουβέντα σε σχέση με τα κοινωνικά θέματα αφορά ουσιαστικά πρώτα-πρώτα την ικανότητα εφαρμογής, υποχρέωσης. Αν τελικά μπορέσουμε αυτά τα στοιχεία της επιβολής δηλαδή και, και τήρησης να τα λάβουμε υπόψη, τότε νομίζω ότι κάτι θα πάει καλύτερα για μας τους αφελείς αισιόδοξους βουλευτές. Έχει το λόγο κύριε για το ΕΛΚ. Φρίλνερ. Πρώτα πρώτα. Μια γενική παρατήρηση. Θεωρώ ότι έχουμε αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το επίπεδο τήρησή του και σεβασμός τους είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το επιλύσουμε. Αυτό όμως δεν είναι λόγος να μην έχουν πολιτικές σχέσεις με μια χώρα. Γιατί άλλο να υπάρχει καταστολή και καταπίεση που είναι κακό, αλλά το να είναι κανείς υποκαταστολή και να είναι και φτωχός αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιηθούν αυτές οι ρήτρες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σαν το καρότο. Όχι σαν μια δικαιολογία αποφυγή συμπορικών σχέσεων, διότι αν δεν υπάρχει εμπόριο υπάρχει φτώχεια και φτώχεια δεν πρόκειται να βοηθήσει την βελτίωση στις επιδόσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ όμως πήρα το λόγο διότι κάτι είπε ο κύριος Ντέβιντ Μάρτιν που μου φέρνει κάτι άλλο στο μυαλό, το διαδίκτυο. Το ίντερνετ σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσο ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ιράν, Μπούρμα, Κίνα, Έγινε αυτό. Και αυτό το οποίο εμένα με ταράζει είναι ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες βοηθούν δικτατορίες. Δικτατορίες να καρβαλίζουν τα δρομένα να κλείσουν το Ιντερνετ, να ξέρω μια σουηδική εταιρεία η οποία ε, με τηλεφωνικό υλικό που χειρίζεται, ε, τηλεφωνική εταιρεία που έδωσε σε μια τρίτη χώρα ονόματα από κάποιους bloggers. Και αυτοί οι bloggers πήγαν φυλακή. Και είναι τώρα κρατούμε συνείδηση επίσης και κάποιες ιταλικές εταιρείε ε, βοηθούν την Κούβα να κάνει λογοκρισία. Νομίζω ότι οι ΙΠΑ το έχουν ψάξει περισσότερο από εμάς. Και έχουμε ένα νομοθέτημα GOFA ονομάζεται στη, στη, στην Αμερική που αφορά ακριβώς αυτό. Αυτό στην αρχή ήταν άσκηση επιχάρτου. Ε, που είχαμε κάνει εμείς εδώ. Δηλαδή, είχαμε προσπαθήσει να δούμε πώς αυτό το νομοθέτημα το αμερικανικό, GOFA, πώς θα το μεταφέρουμε στην Ευρώπη. Δηλαδή, με ένα νομοθέτημα τέτοιο να υποχρεώσουμε τις ευρωπαϊκές εταιρείες να να μην βοηθούν έτσι έμεσα ή στην περιστολή των ελευθεριών. Άρα νομίζω ότι σε αυτό το μέτωπο πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Και γι' αυτό σας λέω ότι επιτέλους για μια φορά ας διδαχθούμε κάτι από τους Αμερικάνους γιατί εκεί τα πάνε καλύτερα. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ο κύριος εκ μέρους της ΕΚΟΕ. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πραγματικότητα είναι ότι πολλοί εδώ θα προτιμούσαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θέματα των διεθνών προτύπων να μην εμπλέκονται καθόλου στα εμπορικά θέματα. Και αυτό ήταν και ο στόχος νομίζω του τελευταίου σχολείου. Δηλαδή να μιλάμε ε, όχι μόνο για ελεύθερο εμπόριο αλλά για εμπόριο χωρίς αξίες με το οποίο εγώ διαφωνώ άρδιν διότι οι άνθρωποι θέλουν να υπάρχει ε, δίκαιη κατανομή και δίκαιοι κανόνες παιχνιδιού για όλους. Πιστεύουμε λοιπόν ότι υπάρχει δυνατότητα να ακούει κανείς την τοπική κοινότητα και ε, να ε, ε, λάβουμε υπόψη μας ότι πολλοί επηρεάζονται από τις πράξεις ορισμένων που ψάχνουν το κέρδος εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέσω μηχανισμών με τους οποίους μπορεί να υπάρχει παραβίαση των αρχών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Κοινοβουλίου των ε, ε, των θεσμικών οργάνων ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και παρόλα αυτά ε, δημιουργούνται ε, συμβάσεις οι οποίες υποβάλλονται για κύρωση. Λοιπόν, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει σε αυτές τις διαδικασίες μέσω των περιπτώσεων που πηγαίνουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο δεν πρέπει να εκπλησόμαστε και τέλος ερχόμαστε στο θέμα του της BP και του δράματος εις τον κόλπο του Μεξικού και ο Επίτροπος είπε ήταν ατύχημα με αυτό τελειώσαμε δηλαδή δεν είναι σωστή αυτή ε, η προσέγγιση για έναν Επίτροπο διότι υπάρχουν ε, σοβαρές ε, αποδείξεις ότι ε, η περικοπή των δαπανών και η επιζήτηση του μεγίστου κέρδους οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση όπως και η περίπτωση της Shell στην Ιγυρία όπου αναφερόμαστε οι θέματα που θίγουν όλη την ανθρωπότητα και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα προβλήματα αυτά θα διορθώσουν Ευχαριστώ. Έφτασε η ώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Λουίς Πορτέρο της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σχολιάσω εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα είμαι πολύ σύντομος. Το πρώτο το οποίο ήθελα να πω είναι το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμμετάσχει στη συζήτηση και σε αυτό το σοβαρό θέμα ε, διότι αναπτύσσουμε την πολιτική και ε, ε, θέλουμε να υπάρχουν ανταλλαγές απόψεων και συνδρομή στα βασικά θέματα. Το δεύτερο πράγμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω εδώ είναι ότι υπάρχει μία διαφοροποίηση μεταξύ συμφερόντων και αξιών και νομίζω ότι ε, υπάρχουν ε, διαφορετικά θέματα μεταξύ των αξιών και ε, των προτύπων διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να προβάλλει τις ευρωπαϊκές αξίες αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να παρακολουθούμε ε, τα οικονομικά συμφέροντα και τις ελάχιστες ε, προδιαγραφές στα διάφορα κράτη διότι εκεί βασίζεται ε, το όλο θέμα. Στις τελευταίες λοιπόν συμφωνίες που διαπραγματεύτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα με την Κορέα προσπαθήσαμε να φτάσουμε εις βάθος και να δούμε πώς εφαρμόζεται η περιβαλλοντολογική νομοθεσία. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να πω ότι βρισκόμαστε σε κεφάλαια τα οποία είναι δεσμευτικά με νομικές δεσμεύσεις και με ένα μείγμα διατάξεων τα κεφάλαια τα οποία διαπραγματεύεται ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα να αναφέρονται εις ε, τη διαδικασία επιλύσεως διαφορών με ανεξάρτητο διαιτητή ο οποίος θα δει ε, κατά πόσον τα μέρη ε, που συνευλήθησαν έχουν σεβαστεί τις προδιαγραφές στο παρελθόν και να διατυπωθούν λύσεις ή να προβλεφθούν κυρώσεις εάν υπάρχει κάποια παραβίαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει από αυτού ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι πιο αποτελεσματικοί για να λύσει κανείς το πρόβλημα αυτό, αλλά θέλουμε να διαχωρίσουμε μεταξύ των ε, ε, ε, των ε, λύσεων και ε, των προβλημάτων. Και υπάρχει και ένα άλλο πολύ βασικό θέμα που είναι η ανάγκη να εξασφαλίσουμε ότι ε, εφαρμόζονται οι διατάξεις και να διασφαλίσουμε ότι ό,τι γράφεται όντως θα εφαρμόζεται και ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να εξασφαλίσουμε τη σωστή παρακολούθηση και εφαρμογή. Είμαι διαθέσιμος για να σχολιάσω περαιτέρω τις τεχνικές ίσως πτυχές που ενδιαφέρουν αυτή την Επιτροπή. Ωραία. Και τώρα η κυρία Σάιφη για να κλείσει το θέμα αυτό monsieur président quelques remarques euh, rapides. d'abord je voudrais remercier les collègues pour leur. Euh, ναι, ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα όσα είπαν και θα ήθελα να επισύρω την προσοχή των συναδέλφων στο ότι αυτή η έκθεση αφορά ανθρώπινα δικαιώματα κοινωνική πρόνοια και περιβάλλον. Δεν θέλουμε να υπάρχει άνηση αντιμετώπιση. Είναι σημαντικά τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα θέλουμε επίσης να προσέξουμε επίσης. Όχι, δεν θέλουμε όλα αυτά να μείνουν καλές προθέσεις, θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Ρεαλιστές και να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτό το θέμα. Όχι, δεν θέλουμε με αφέλεια να προσπαθούμε να πετύχουμε τόσα πολλά που τελικά τίποτα δεν πετυχαίνουμε. Ε, πάνω σε αυτό θα λάβω υπόψη αυτό το οποίο είπατε. Μάλλον και πιστεύω ότι όντω οι πολιτικέ πτέρυγε του Κοινοβουλίου πρόκειται να καταφέρουν την συνένεση, διότι νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε ε, ακόμα και με μικρά βήματα, αλλά να προχωρήσουμε. Αυτά και ευχαριστώ την Κομισιόν για τα όσα είπε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρο. Σα υπενθυμίζω ότι η εξέταση θα γίνει στι 28 Ενάτου. Έχουμε ήδη λάβει τις γνωμοδοτήσεις από τις συναρμόδιες επιτροπέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβάλλοντος. Το επόμενο. Εμπορικές σχέσεις ΕΕ με Λατινική Αμερική. Έχουμε ένα εγγραφό εργασία το οποίο συνετάγει από τον εισηγητή Helmut Scholz, τον συνάδελφο της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς. Όπως γνωρίζετε, έχουμε κάποιες πρόσφατες εξελίξεις στην Λατινική Αμερική. Έχουμε κάποιες διαπραγματεύσεις που είχαν κάποια αίσια κατάληξη. Περού, Μερκοσούρ και η Επιτροπή μας παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις εν ενός νέου πλαισίου μερικών σχέσεων με την Λατινική Αμερική. Επομένως, είναι πολύ σημαντική έκθεση τούτη. Γι' αυτό και θα δώσω το αντισκητάλι στον Helmut Scholz για να παρουσιάσει το έγγραφο εργασία που συνέταξε. Ευχαριστώ. Καταρχήν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 η Επιτροπή μου ανέθεσε την, το έργο να κάνω μία έκθεση κατά πρωτοβουλία για το θέμα των εμπορικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσης με τη Λατινική Αμερική για να εξετάσουμε ε, διάφορες πτυχές οι οποίες μας απασχολούν. Ε, ήδη θεωρούμε ότι το θέμα αυτό είναι πολύ επίκαιρο και με την έκτη διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ενώσεως Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής στη Μαδρίτη έχουν διαγραφεί τα, οι βασικές αρχές των εμπορικών σχέσεων και εάν θέλουμε να εξετάσουμε τις εμπορικές σχέσεις θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την προϋπόθεση ότι πρέπει καταρχήν να στραφούμε προς τις προοπτικές για το μέλλον ε, όπως σας έχω πει υπήρξε μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων και εκεί είχα θέσει διάφορα ερωτήματα. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τρόπον ώστε να θέσει τις ε, ε, τις ε, σχέσεις σε ένα γενικό πλαίσιο και να εξετάσει τις ιστορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ των Ευρω... της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Λατινικής Αμερικής. Τι μπορούμε δηλαδή να κάνουμε κατά τρόπον ώστε ε, το εμπόριο αυτό να εξασφαλίσει την ε, ευημερία ε, των ανθρώπων στις χώρες αυτές και να μπορέσει να επηρεάσει θετικά και να προωθήσει τα άτομα και τους ανθρώπους στην περιοχή. Ε, είπαμε ότι έπρεπε να γίνει ε, επίσης ε, μία μια εξέταση των ανθρώπων στις χώρες αυτές κατά τρόπον ώστε να εξετάσουμε την περιφερειακή την ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας έγινε μια ενδιαφέρουσα ακρόαση όπου μιλήσαμε με τους υπευθύνους των περιοχών δηλαδή Κεντρικής Αμερικής ε, Ειρηνικού αλλά συγχρόνως και Μεξικού και Κίνας για να μπορέσουμε να αναλύσουμε τα θέματα αυτά και στο έγγραφο εργασίας προσπάθησα να διαγράψω μία συγκεκριμένη κατεύθυνση να δω κατά πόσον είναι ε, ισοσκελισμένες οι σχέσεις οι εμπορικές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ε, Λατινικής Αμερικής ε, πόσο η διάσκεψη κορυφής ασχολήθηκε ε, με τις εξωτερικές σχέσεις και στα πλαίσια της Επιτροπής μας να εξετάσουμε το περίπλοκο θέμα της, ε, του εμπορίου ε, ανάπτυξης και προώθησης κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε ε, να βελτιώσουμε τις ε, πολυπληθείς ε, διεργασίες οι οποίες γίνονται στην περιοχή αυτή. Ξέρουμε ότι είναι πολύ περίπλοκο το θέμα, το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως εδώ, άρα ο κύκλος των προβλημάτων για την κατάσταση μεταξύ Περού και Βολιβία όπως επίσης και το πρόβλημα του Ισημερινού, το πρόβλημα του εμπορίου της μπανάνας, ε, το προβλήματα των χωρών και της Καραϊβικής, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία είναι σημαντικά για το εμπόριο και θα έπρεπε να τα εξετάσουμε πιο συγκεκριμένα. Στο τέλος λοιπόν της ομιλίας μου ε, αναφέρθηκε αναφέρθηκα σε ορισμένα θέματα ή ορισμένες διατυπώσεις ε, διατυπώσεις οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε εδώ ένα πρώτο σχέδιο της εκθέσεως αυτής ε, θα μπορούσαμε ίσως να συζητήσουμε τα θέματα αυτά προτού προχωρήσουμε σε ένα έγγραφο εργασίες για να έχουμε συμφωνήσει ως προς το τι χρειάζεται να γίνει. Επίσης θα πρότεινα να υπάρχει ένας ε, σκιώδης εισηγητής και να είμαστε σε στενή συνεργασία κατά τρόπον ώστε να συζητάμε ευθύ εξ αρχής το σχέδιο που θα καταρτήσω μαζί και να μπορέσουμε από κοινού ε, να παρακολουθήσουμε την διαμόρφωση της εκθέσεως μέχρι το τέλος της. Και επίσης από πλευράς χρονοδιαγράμματος όπως σας είπα προσπαθούμε ε, να συζητήσουμε το σχέδιο αυτό στην συνεδρίασή μας του Ιουλίου στην Επιτροπή μας και τον Οκτώβριο να υποβληθεί για ε, ψηφοφορία η συνολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και προσβλέπω στην βελτίωση και ανάπτυξη αυτού του εγγράφου. Ευχαριστούμε κύριε Σόλτ. Το χρονοδιάγραμμα είναι αυτό που είπατε κι εσείς. Εξέταση της εκθεσής σας στην συνάντηση του Ιουλίου. Και καλό τα μέλη της Επιτροπής μας να μας αποστείλουν τα σχόλια τους για το σχέδιο του κειμένου. Ιδίως τα σημεία που επισημάνατε κι εσείς. Αυτό που έχετε συμπεριλάβει στο τελικό μέρος του εγγράφου σας. Ο κύριος Κάζακ από την άλλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Βρίσκω ότι το έγγραφο εργασία που ετέμισε ο κ. Σόλτ είναι διεξοδικό, καλύπτει πολλέ πτυχέ των σχέσεων με τη Λατινική Αμερική και ακόμη και αν δεν συμφωνώ με όλες τι θέσει που εκφράζονται στο έγγραφο, θεωρώ ότι είναι διεξοδική η εξέταση του θέματος και πολύ καλή επισκόπηση. Νομίζω ότι η σύνοδος που οργανώθηκε το 2008 στη Λίμα με τις χώρες της ε, ΑΚΕ ήταν ε, πολύ θετικές για να ορίσουμε τις εταιρικέ μας σχέσεις με τις χώρες αυτές. Ο εισηγητής ε, ανέφερε κάποιες πρόσφατες εξελίξεις, όπως η λύση που προτάθηκε για το εμπόριο της μπανάνας στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Ωστόσο, απομένουν πράγματα που πρέπει, στοιχεία που πρέπει να αποσαφινιστούν. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι ασιατικές χώρες ανταγωνίζονται μαζί μας στο πεδίο της Λατινικής Αμερικής. Αυτό επαριλημμένως αναφέρεται στο κείμενο του κ. Σόλτς και σίγουρα περισσότερα βιομηχανικά προϊόντα πολλούμε στην Νότια Αμερική παρότι βασικά προϊόντα εισάγουμε. Το αναφέρει συχνά ο συγκεκριτή στο κείμενο τους στόχους της χιλιετίας του ΟΗΕ και είμαι της άποψης ότι το εμπόριο θα μπορούσε να διευκολύνει την επίτευξη αυτών των στόχων, οπωσδήποτε, χωρίς όμως να επικρίνουμε κι εμείς τόσο σφοδρά τις ε, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Ίσα ίσα που νομίζω θα μπορούσαν να είναι ευεργετικέ και να διευκολύνουν την επίτευξη των στόχων. Επίσης, ο κ. Σόλτ υπογραμμίζει τις διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ και την διαπραγματευτική εντολή εκεί θα χρησιμοποιηθεί. Εγώ, συζητώντα με τον Επίτροπο Δεκούκτ, είχα την εντύπωση ότι δεν είναι πλήρω διτεθειμένο να αναθεωρήσει ή να τροποποιήσει την διαπραγματευτική εντολή τη Επιτροπή. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιε θα είναι οι εξέλιξει σχετικά. Επίση, υπάρχουν πολλέ συστάσει στο έγγραφο εργασία για την πλευρά της ανάπτυξης. Είναι σημαντικά στοιχεία μεν, αλλά πιστεύω ότι περισσότερο έπρεπε τη αρμοδιότητα τη επιτροπή ε, Ανάπτυξης, ΔΕΒΕ, του Κοινοβουλίου, παρά τη δική μα επιτροπή. Επίσης είμαι τη άποψη ότι η οικονομική εξάρτηση πρέπει να αποφεύγεται, φυσικά, αλλά θα απέφευγα διαπιστώσεις κάπως βιαστικές χωρίς να περιμένουμε να δούμε τι θα δώσει η συνέχεια της εμβάθυνσης των σχέσεων μας με τη Λατινική Αμερική. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν θα παρακολουθήσω τη συνέχεια της συζήτησης. Μου φαίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη και επικοδομητική για όλους μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Άλμπα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Σόλτς για την έκθεση του. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλή η παρουσίαση που, που γίνεται στην έκθεση. Παρόλα αυτά, δεν θα ήθελα να σταθώ στα θετικά σημεία της έκθεσης. Θα συμφωνήσω με τον εισηγητή ε, ως προς το ότι το εμπόριο και τα εμπορικά εργαλεία, τα μέσα, είναι ένα επιπλέον εργαλείο για να καταπολεμήσουμε την ε, οικονομική κρίση την οποία διανύουμε. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα πρέπει να ενισχύσουμε όλα τα μέσα που επιτρέπουν την περαιτέρω αναθέρμανση του εμπορίου, όπως τις εξαγωγές και βεβαίως τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον, η υγεία οι κοινωνικέ διαστάσεις είναι θέματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Το εμπόριο, πιστεύω, μπορεί να είναι και ένας μηχανισμός προόδου, ολοκλήρωσης. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε όλα τα διατηθέμενα μέσα και για τους παραγωγούς και γεωργούς μας, γιατί είναι ευκαιρία οι μεγάλες επιχειρήσεις και εταιρείε κατά την υπογραφή μια συμφωνία με τρίτη χώρα ή ε, τρίτη μια γεωγραφική ζώνη εκτό Ευρώπη να υποφελούνται. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα προϊόντα που μπορούν να εξάγονται και νομίζω η εμβάθυνση των εμπορικών σχέσεων θα επιτρέψει τις δυσαναλογίες που υπάρχουν ως προς τις εισαγωγές και εξαγωγές να τις καλύψουμε και να στραφούμε από κοινού με τις τρίτες χώρες σε τομείς πιο παραγωγικούς για τις σχέσεις με την κοινότητα των Άνδεων και στο πλαίσιο με τη συμφωνίας με την Κολομβία και το Περού η συμφωνία αυτή προφανώς έχει πολλές, μετα... πολλές συγκεκριμένες ρήτρες που αφορούν το Περού και ίσως και την κοινότητα των Άντζων κατ' επέκταση και αυτό θα είναι και η βάση μας με ολόκληρη αυτή τη γεωγραφική περιοχή και γενικότερα την, Αμε... την Λατινική Αμερική. Αυτό θα μας φέρει πιο κοντά με τις δύο αυτές χώρες που θέλουν να προχωρήσουν στις σχέσεις μας. Ο Ισημερινός τώρα ίσως να κάνει το ίδιο σε ένα προσεχές μέλλον. Ίσως να αναλυφθούν ε, ξεχωριστές πρωτοβουλίες, να μην συμμετάσχει στην ομάδα των άλλων χωρών δηλαδή, για πολιτικούς λόγους, όμως η πρόοδος των σχέσεών μας με τις άλλες χώρες είναι κάτι που το βλέπουμε ο καθένας από διαφορετική σκοπιά. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση όμω να πάψουμε τι προσπάθειε. σα ίσα θα πρέπει να τι εντείνουμε. Για τη Μαρκοσούρ θα πρέπει να προσπαθήσουμε να σταθεροποιήσουμε τι σχέσει μα. Έχουμε πολεμήσει για μια ισορροπή συμφωνία η οποία να ωφελεί και τι δύο συμβαλλόμενε πλευρέ, και τι χώρε τη Μαρκοσούρ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα το Ευρωκοινοβούλιο, συμφωνώ μαζί σα, πρέπει στενά να παρακολουθεί και να συμμετέχει ενεργά στι διαπραγματεύσει αυτέ. Πρέπει επίση να έχουμε υπόψη ότι ο πρόεδρο Διακόπτε τον ομιλητή. Οι συμφωνίε αυτέ είναι συμφωνίε που πρέπει οπωσδήποτε να υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριο Μενέντε, από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, συμφωνώ με τη γενική φιλοσοφία της έκθεσης που μας υπέβαλε ο συνάδελφος Σόλτς. Συμφωνώ λοιπόν μαζί του και συμφωνώ με τα γενικότερα αισθήματα που υποκίνησαν αυτή τη γενική φιλοσοφία του. Υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία συμφωνούμε και άλλα στα οποία προφανώ διαφωνούμε και αυτά θα ήθελα να σχολιάσω. Είναι σαφέ και το λέω προκειμένου να συντομεύσω ε, και θέλω να είμαι σύντομο ευθύ εξ αρχή ότι όποιος δεν, ποιος δεν θα μπορούσε μάλλον να, συμφωνήσει με τον κύριο Σόλτ όταν λέει ότι η Λατινική Αμερική θα εξασφαλίσει την ε, ευημερία της χάρη στο εμπόριο. Ναι, λέει ότι το να δίδονται πλεονεκτήματα με τρόπο ισότιμο είναι σίγουρα είναι κάτι θετικό. Πώς να μην συμφωνήσουμε επίσης όταν ε, λέει ότι η διμερής πρόοδος, η εξέλιξη δεν θα πρέπει να εξωθήσει τους εταίρους να εγκαταλείψουν τους διμερείς στόχους τους. Ε, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Υπάρχουν διμερεί στόχοι. Στόχοι που δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα τους εγκαταλείπουμε όποτε περνάμε σε πολυμερείς διαπραγματεύσεις. Και πώς να μην αναγνωρίσουμε ότι είναι απαραίτητη η σύναψη συμφωνίας της Δόχα η οποία να είναι δίκαιη και να επιτρέπει ίσες ευκαιρίες καταπολέμησης της φτώχειας στη Λατινική Αμερική. Όλα αυτά είναι ορθότατα. Συγχαρητήρια. Μπράβο σας. Η ε, ανάλυση του θέματος είναι πολύ σωστή. Να διευκρινίσω εδώ, μιας και μιλάτε για τα εμπορικά ωφέλη, ότι δεν θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ του βαθμού ανάπτυξης ε, μετα... όπως της Βραζιλίας και της Βολιβίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη συγκρίνοντας αυτές τις δύο χώρες μεταξύ τους, διότι οι αναπτυξιακές τους διαφορές είναι αξιοσημείωτες. Επίσης, η Ένωση συμβάλλει δυστυχώς ε, τα μέγιστα στην ανάπτυξη με την βοήθεια, την αναπτυξιακή της βοήθεια και με το σύστημα Aid for Trade, βοήθεια για το εμπόριο. Ίσως θα ήταν καλό να εντείνουμε τις προσπάθειες συντονισμού και τις ε, κινήσεις ευρωπαϊκής βοήθειας. Εδώ δεν ήθελα να μακρηγορήσω, ήθελα απλώ να σταθώ σε αυτά τα τρία σημεία τα οποία βρίσκονται σε σημεία απόκληση σε σχέση με την τοποθέτηση του κυρίου Σόλτ. Ε, και να θίξω το βασικό θέμα που έθιξε και ο συνάδελφο. Ούτε η πολιτική μα ομάδα να δεχτεί το ότι άπαξ και η Βολιβία δεν αποσύρει αυτό το αίτημα Δηλαδή αυτό το δικαστήριο της ε, κοινότητας των Άνδεων δεν ε, ανατρέπει αυτό το αίτημα της ε, Βολιβίας ότι θα πρέπει να παγώσουμε τις σχέσεις. Δηλαδή δεν θα πρέπει εμείς να καταστούμε όμοιροι της δικαστικής αυτής απόφασης. Πάντως πολύ καλά τα ο Σάλβα ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποια νέα, κάποια νέα αξιόπιστα ότι δηλαδή πρόκειται η Βολιβία να αποσύρει αυτή τη την προσφυγή του αίτημα ίσα το, το δικαστικό αυτό όργανο και επίσης ε, έχουν υπάρξει κάποιες ε, ε, κινήσεις τις τελευταίες μέρες σε σχέση με το ότι η Βολιβία είναι διατεθαμένη να μην είναι σε σχέση με το Εκουαδόρ και ότι θέλει να προσυπογράψει τη λεγόμενη συμφωνία ανάπτυξης. Έχουμε αυτά τα banana company μέσω στα 200 εκατομμύρια ευρώ, που μας παρέχουν εγγύσεις προς την επιθυμία κατεύθυνση. Επίσης, τρίτο και τελευταίο για το Mercosur, εκτός από την Κομισιόν και τον κύριο Ντεχούχτ. Δεν σημαίνει αυτό θα περάσει ό,τι θέλουν και εμείς μπορούμε να είμαστε και δηλαδή ότι δηλαδή έχουμε αυτή την ε, δεκαετία που θα, ε, θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Γιατί μπορεί με να έχουμε αυτή την παγκοσμιοποίηση και τη σχετική αντιμετώπιση, αλλά θα πρέπει να δούμε πρώτα-πρώτα τι θα κάνει ο Μερκοσούρ. Και άλλα πολλά μπορώ να σας πω. Αλλά μια που δεν λέγομαι τη δεν μπορώ να, να πω περισσότερα. Πρέπει τώρα να βάλω τελεία. Ε, καλά πρώτη συζήτηση είναι του, του, του σχεδίου εγγράφου, λέει ο Πρόεδρος. Θα τα ξαναπούμε, να, τον Ιούλιο κιόλας. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος ε, Ματίας Γιώργης είναι έχει το λόγο. Σύντομα παρακαλώ. Κάποια σύντομα σχόλια έχω πρόεδρε. Με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά των σχέσεων μας με την Λατινική Αμερική. Πολύ καιρό θέλατε να συσφίξουμε σχέση με την Λατινική Αμερική στο παρελθόν και επίσης Άρα γι' αυτό μας χαροποιεί το ότι συνεχίζεται να δείχνει τέτοια στάση. Εμεί συμφωνούμε με τα περισσότερα που αναφέρονται στο σχέδιο τη έκθεση. Νομίζω ότι συγκλίνουν οι απόψεις μα. Και όπω λέει και η έκθεση, θα πρέπει μέσω των συμφωνιών αυτών να προωθήσουμε εμπόριο, επενδύσεις, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει στο γενικότερο πλαίσιο των σχέσεων που θέλουμε να χτίσουμε τη Λατινική Αμερική. Δηλαδή, να προωθήσουμε κοινωνική συνοχή, περιφερειακή ολοκλήρωση, ε, ανάπτυξη αηφόρο και τους απτυσιακούς στόχους της χιλιετίας. Γι' αυτό και συνάπτουμε τέτοιε συμφωνίε που δεν είναι μόνο συμφωνίες ελευθερών να αλλά και συμφωνίε σύνδεσης, συνεργασία και πολιτικού διαλόγου. Όντω πρέπει και οι δύο πλευρέ να είναι λογικές στα αιτήματά τους, να έχουμε σταδιακή απορρίθμιση. ευελιξία, επίοικια, συνοδευτικά μέτρα, ενδυνάμωση των θεσμικών φορέων εξαγωγών και εισαγωγών και έτσι νομίζουμε θα χτίσουμε πιο στενούς με τη Λατινική Αμερική. Τέλος. ένα σημείο στο οποίο διαφωνούμε. Αναφέρθηκε η Βολιβία και συμφωνούμε με το ότι αυτή η διαφορά η το των δικαστηρίων είναι εσωτερικό θέμα. Αλλά όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Βολιβία είναι η πιο ευεργετημένη από τις επιλέξιμες χώρες για να η βοήθεια στην Νότια Αμερική. Να προσαρμόσουμε βεβαίω τι σχετικέ οδηγίε για τι διαπραγματεύσεις, Αλλά δεν είναι ότι αυτό είναι αναγκαστικά η μόνη οδός. Δεν θέλουμε ούτε να υπάρχει ένα απομόνωση. έχουμε και παρελθόν, θα έχουμε και μέλλον σε τέτοιου είδου πολιτική. Πάντω, ε, εμεί ευχαριστούμε να ακούσουμε απόψει και να τι λάβουμε υπόψη. Και να σημειωθεί πρόοδο στι διαπραγματεύσει. Αλλά κυρίω εκτιμούμε το πόσο ενδιαφέρεστε. Και είναι πάρα πολύ θετικό το ότι συμφωνούμε σε αυτή την πολιτική που θέλουμε να χαράξουμε και που ξεκίνησε από τη συνάντηση του Μαΐου της Μαδρίτης. Θέλω να δευτερολογήσει ο εισηγητής μας, ο κύριος Χέλμουτ Σόλτς. Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος διότι ε, ε, ε, συμφωνώ ότι ενδέχεται να υπάρχουν διγνωμίες και σημεία στα οποία δεν συμφωνούμε. Όταν μιλάμε όμως για αυτές τις εμπορικές σχέσεις ειλικρινά θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο συγκεκριμένο θέμα το οποίο συζητάμε και είχα την ευκαιρία στους τελευταίους μήνες και εβδομάδες να επισκεφθώ ορισμένες χώρες στην περιοχή να συζητήσω με ε, τα άτομα τα οποία επηρεάζονται από το διεθνές εμπόριο και το τι περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τρόπον ώστε να, να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν και προσδοκίες αλλά και υπάρχει ο φόβος ότι οι χώρες αυτές ε, με τις οποίες συναλλασσόμαστε μπορεί ε, να κλείσουν και θα πρέπει να γίνει μία ανταλλαγή επίσης βάσεως να γνωρίζουμε τον ε, ε, συμβαλόμενό μας ε, με τον ίδιο τρόπο και γι' αυτό είπα ότι το, στις συμφωνίες Μερκοσούρ τώρα το, η Βραζιλία είναι ε, μια χώρα με μεγάλη αυτοπεποίθηση και λένε αν δεν μας πάρετε στα σοβαρά θα διαπραγματευτούμε με άλλους. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιληφθεί ότι πρόκειται για μια νέα πρόκληση την οποία να αντιμετωπίζουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά κάποιον τρόπο πρέπει να υπάρξει μια αμοιβαία ανταλλαγή κατά τρόπον ώστε να σκεφτούμε πώς θα οργανωθούμε. Το τρίτο θέμα που με ενδιέφερε ήταν ότι με ενδιέφερε πάρα πολύ η μακροπρόθεσμη στρατηγική η οποία συζητήθηκε σήμερα με τον κύριο Ντεγκούχτ διότι πιστεύω ότι τώρα μας δίδεται η ευκαιρία να περιλάβουμε και αυτόν τον στρατηγικό προσανατολισμό ή την προσέγγιση μας για το πόσο θα διοργανωθούμε και θα διοργανώσουμε τις συνεργασίες μας ιδίως με αυτές τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει ε, καταρχήν ε, να ε, παρουσιάσουμε το σχέδιο ε, εκθέσεως και να δούμε ε, πώς θα διαπραγματευτούμε με τις χώρες αυτές όπως και στον Ισημερινό όπου είναι θέμα ζωής και θανάτου. Εάν έχουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά αυτό συμβαίνει ότι θα πρέπει και εμείς και η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είμαστε πολύ ευαίσθητοι για το πώς θα οργανωθούμε για να μην υπάρξουν αντιπαλότητες αλλά για να οικοδομήσουμε αυτή τη σχέση και να περιλάβουμε και τους παραγωγούς και ε, τους ε, ε, εμπόρους για τις μπανάνες. Υπάρχει σχέση στα πλαίσια του ΠΟΕ και η σχετική ρύθμιση, άρα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε αυτά να τα συνδυάσουμε και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο και πιστεύω ότι θα έχουμε ε, μία πολύ στενή συνεργασία κατά την κατάρτιση του εγγράφου για να μπορέσουμε να δώσουμε δυνατότητε στις χώρες αυτές. Θα περιμένουμε το σχέδιο έκθεσης και θα το συζητήσουμε στη συνάντηση του Ιουλίου. Σας ευχαριστώ όλους και περνάμε στο σημείο 15. Διαπραγματεύσεις για Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας και σχετικές διαπραγματεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά με την Ινδία στις διαπραγματεύσεις αυτές για θέματα προϊόντων και υπηρεσιών. Είναι διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν από το 2007. Οκτώ διαπραγματευτικοί γύροι έχουν λάβει χώρα ως τώρα και ο πιο πρόσφατος έλαβε χώρα στο Δελχή τον Ιανουάριο φέτος. Η Ινδία, όπως ξέρετε, είναι σημαντικότατος εμπορικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση με αυξηνο... και αυξανόμενη οικονομική δύναμη. Με πληθυσμό περισσότερο του ενός δις 200 εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία στον κόσμο ή μεταξύ των ταχύτερων. παρακολουθούμε στενά τις διαπραγματεύσεις αυτές και νομίζω ότι είναι επίκαιρο να κάνουμε τώρα μια ανταλλαγή απόψεων για το συγκεκριμένο θέμα, για το πώς έχουν προχωρήσει ως τώρα οι διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Επιτροπή, στον ε, κύριο Γκνάθιο Γκαρσία. Έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε, είναι μεγάλη μου χαρά που έχω την ευκαιρία να σας δώσω μια επισκόπηση για το που έχουν φτάσει οι διαπραγματεύσει μας με την Ινδία. Όπως σωστά επισημάνατε, αυτή είναι μια σοβαρότατη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον περατώσουμε τη συμφωνία με την Ινδία. Κάτι που είναι αρκετά φιλόδοξο και αν έχουμε μια τέτοια συνολική συμφωνία θα έχουμε δυνατότητα να περάσουμε σε μια πολύ ταχύως αναπτυσσόμενη αγορά. Τώρα να δούμε γιατί έχουμε φτάσει σε κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων. και αν θα μπορέσουμε να επιλύσουμε κάποια από τα βασικά σημεία, τα βασικά προσκόμματα που μας έχουν εμποδίσει από εδώ να περατώσουμε τις διαπραγματεύσεις αυτές. Η εντύπωση μου είναι ότι η Ινδία αυτή τη στιγμή έχει ενεργό πλέον συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις, συνειδητοποιεί ότι εφόσον η συμφωνία αυτή συναυθεί θα πρέπει να ληφθούν και κάποιε δυσχερεί πολιτικέ αποφάσει από τη δική του πλευρά και το θέμα είναι αν θα υπάρξει προθυμία να τα εξετάσουν τα ζητήματα αυτά. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σα παρουσιάσω όλε τι λεπτομέρειε. Απλώ να τονίσω τρία ζητήματα κατεξοχήν οικονομικά και όπου η πρόοδο ε, η οποία θα επιτελεστεί θα είναι καθοριστική για το πώ θα εξελιχθούν και οι διαπραγματεύσει να τα φτάσουν στο τελικό του στάδιο. Το πρώτο είναι οι δασμοί. Η Ινδία έχει κάνει μια πρώτη προσφορά για τους δασμούς, αρκετά ενδιαφέρουσα, η οποία εξαλείφει τους δασμούς στο 90% των βορευωμένων ειδών και δασμολογικών γραμμών. Όμως θέλουμε κι άλλο ε, κι άλλα ανταλλάγματα από την Ινδία. Κυρίως θέλουμε να βελτιώσει την προσφορά της η Ινδία σε έναν αριθμό καθοριστικών οικονομικών κλάδων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, τα κλωστεφαντουργικά, τα χημικά προϊόντα, οι μηχανικοί εξοπλισμοί και κάποια γεωργικά προϊόντα. Έχουμε καταστήσει σαφές στους Ινδούς συναδέλφους ότι αυτό είναι μια αυστηρή επιταγή. Η Ινδία να συμπεριλάβει κάτι παραπάνω στην προσφορά τη. Εάν μετακινηθεί από την αρχική τη θέση όμω η Ινδία και εμεί το ίδιο θα κάνουμε και τελικά ίσω να μπορέσουμε να εξαλείψουμε δασμού από ό,τι σκοπεύει να το κάνει η Ινδία. Όμω οι δασμοί θα είναι ένα από τα κρίσιμα σημεία όπου θα κρυθούν οι διαπραγματεύσει. Το δεύτερο σημείο είναι οι υπηρεσίες. Η Ινδία είναι ένα ενεργότατο ε, συνομιλητή μα στις διαπραγματεύσει τη Γενέφη. Είναι από τι χώρε που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τι υπηρεσίε, στα πλαίσια των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, όμω το πλαίσιο αυτών των διμερών γύρων. Ελπίζουμε η Ινδία να ξεπεράσει τις προτάσεις που έκανε στη Γενέβη. Εδώ θα πρέπει να συμπεριληφθούν τομείς οικονομικής σημασίας, ευαίσθητοι όπως οι ασφάλειες, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και η λιανική πώληση. Αλλά είμαστε σαφείς, εάν η Ινδία κάνει κάποια παραχώρηση και εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παραχωρήσουμε κάτι. Και η δική μας τάση θα είναι επίσης καθοριστική σημασία για τις διπλωματεύσεις. Η προσωρινή επίσης ε, μετακίνηση Ινδών επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες θα είναι ένα γεγονός που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δεν μιλάμε εδώ για μαζική μετανάστευση, αλλά για προσωρινή μετακίνηση Ινδών με άριστες δεξιότητες που μπορεί να χρειαστεί να πουλήσουν σε εμά υπηρεσίες τους. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε και εμεί την ίδια πολιτική ευαισθησία που απαιτούμε από εκείνου. Το τρίτο σημείο που είναι σημαντικό από εμπορική άποψη και θα είναι καθοριστικό για του ερχόμενου μήνε είναι οι δημόσιοι διαγωνισμοί. Εδώ ξέρουμε ότι θέλουμε να ανοίξουν οι αγορέ των διαγωνισμών, των προμηθειών. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που προωθούμε σε όλε μα τι ε, εμπορικέ διαπραγματεύσει και για την ώρα η Ινδία δεν έχει εντολή να διαπραγματευτεί για το θέμα αυτό. Όμω έχουμε ξεκαθαρίσει ότι το σημείο αυτό για μα θα είναι αποφασιστικό για την εξέλιξη τη συμφωνία. Ελπίζω ότι του προσεχεί μήνε ε, θα έχουμε κάποιε πολιτικέ αποφάσει και σε αυτά τα ζητήματα. Προφανώ θα περάσουμε από κάποια δύσκολα στάδια. Ένα ζήτημα που αναμένουμε να μα δυσκολέψει με την Ινδία είναι το εμπόριο και η βιώσιμη ανάπτυξη. Ήδη έχουμε εξηγήσει στους Ινδούς ότι αυτό είναι ύψης της για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του λόγου. Επίση, σημαντικό είναι να καταστήσουμε σαφέ ότι μεταξύ του σημερινή μέρα και του Οκτωβρίου θα έχουμε τη Σύνοδο Κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση Ινδία. Θα είμαστε σε στενή συνεργασία και επαφή με του Ινδού συναδέλφου για να διερευνήσουμε πού ενδεχομένω θα καταφέρουμε να πετύχουμε πολιτικές ριζικές λύσεις για όλα αυτά τα ζητήματα. Εάν τα ζητήματα αυτά διευθυνθούν από τώρα στον Οκτώβριο, τότε πραγματικά θα υπάρχουν σοβαρέ ευκαιρίε οι διαπραγματεύσει να περάσουν στο τελικό του στάδιο και ενδεχομένω η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών να περατωθεί ω το δυνατόν συντομότερα μετά τη Σύνοδο του Οκτωβρίου. Αυτό όμω θα απαιτήσει την ενεργό συμμετοχή και τι εντατικέ συζητήσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των ε, συναδέλφων μας από το Υπουργείο Εμπορίου της Ινδίας. Αυτό σημαίνει ότι και στο επίπεδο των επικεφαλής διπραγματευτών ε, και στο επίπεδο όλων των συμμετεχόντων θα υπάρχει πολύ σοβαρή αφοσίωση στο σκοπό μας. Πάντως οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι πολύ σοβαρές και γι' αυτό καλωσορίζουμε οποιαδήποτε ερώτηση, απορία μπορεί να έχει το Ευρωκοινοβούλιο είτε για τα ζητήματα που ανέφερε είτε για οποιαδήποτε πτυχή των διαπραγματεύσεων. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Σημειώνω ότι ο συνάδελφος, ο κ. Βότσον, που είναι πρόεδρος της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας, είναι μαζί μας. Τον καλωσορίζω και τον ρωτώ εάν θέλει να ξεκινήσει εκείνο τη σειρά των ερωτήσεων και να συμμεριστεί τις απόψεις του μαζί μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, αυτή είναι η πρώτη ευκαιρία που είχα να παρακολουθήσω τις συζητήσεις της Επιτροπής σας ε, στη διάρκεια αυτής της θητείας και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον άκουσα τα όσα είπατε υπό το σημείο 13 με την αφορμή την έκθεση της κυρίας Σαΐφη. Εκεί εκφράζεται η άποψη ότι το Κοινοβούλιο χρειάζεται περισσότερο εντελεχείς συζητήσεις για την σύναψη τέτοιων συμφωνιών. Ο κύριος Higgins ε, πεσήμανε τα διάφορα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, τα οποία βεβαίως και ε, είναι εύστοχο εδώ να αναφέρονται. Όμω θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ των διαφόρων καθεστώτων και των δημοκρατικών πολιτευμάτων που ενδεχομένω να έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Η Ινδία νομίζω δεν είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η Ινδία έχει 2% μερίδιο τη αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εμεί έχουμε 17% μόνο ε, μερίδιο στη δική του. Ε, είναι λοιπόν ε, εφικτό και προ όφελο και των δύο πλευρών να επεκταθούν οι εμπορικέ μα σχέσει. Νομίζω μάλιστα ότι θα ωφελήσει λίγο περισσότερο εμάς ως προς τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι επιχειρηματικές μας δυνατότητες ανάπτυξης στη χώρα αυτή. Πάντως το μήνυμα που έλαβε η αντιπροσωπεία μου μιλώντας μετά τους, με τους Ινδούς υπουργούς και τους Ινδούς νομοθέτες είναι ότι ενδιαφέρονται για μια συμφωνία μαζί μα, αλλά όχι για συμφωνία που να ξεπερνά τα εμπορικά ζητήματα. αυτό είναι κατηγορηματική. Στο πλαίσιο τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών είναι πρόθυμοι να συζητήσουν και άλλα ζητήματα. Αλλά σε άλλα φόρουμ, αν θέλουμε εμπορική συμφωνία, ε, μα λένε ότι θέλουμε να περιορίζεται στα εμπορικά ζητήματα. Αυτό μα φέρνει στην εξή θέση. Ή δεν θα έχουμε καθόλου συμφωνία, Οπότε θα στερήσουμε από του δικού μα πολίτε και του Ινδού πολίτε, από τα, τα ωφέλη, τα ευεργετήματα μια τέτοια συμφωνία ή θα αποφασίσουμε να προχωρήσουμε στην πορεία τη συμφωνία αυτή, αλλά σε άλλο πλαίσιο, δηλαδή ενδεχομένω να μην συζητήσουμε μαζί του κοινωνικά και, και περιβαλλοντικά ζητήματα. Εγώ πιστεύω ότι αν μας απασχολούν τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στην Ινδία, πράγμα που σωστό είναι, θα πρέπει να διερωτηθούμε το εξής. Είναι καλύτερο να επιδιώξουμε το σεβασμό των προτύπων αυτών με μια αμοιβαίω ωφέλιμη εμπορική συμφωνία που να συνοδεύεται και από συζητήσει άλλα ενδεχομένω πλαίσια και φόρα ή να περιοριστούμε στο εμπόριο. Θα έχουμε περισσότερη δυνατότητα πίεση από ό,τι τώρα. Επιζητούμε μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών από το 2006 με την Ινδία. Οι εξαγωγεί μα συνεχώ αντιμετωπίζουν καταστάσει όπου, όπου τα 28 διαφορετικά κράτη τη Ινδία λαμβάνουν αποφάσει που επηρεάζουν το εμπόριο και επιφέρουν σοβαρότατο κόστο στι διάφορε εμπορευόμενε εταιρείε. Νομίζω λοιπόν πολλοί από εμά σε αυτό το σώμα θα προτιμούσαν μια πολυμερή εμπορική συμφωνία στο επίπεδο τη Δόχα. Αλλά εφόσον κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί, τότε η αντιπροσωπεία μα θα θεωρού, θεωρεί μάλλον ότι θα είχε σοβαρά ωφέλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών πρόεδρε, όταν πήγαμε στην Ινδία, συναντήσαμε και του αντιρρησίε από την πλευρά των Ινδών σε σχέση με μια συμφωνία ελευθερου εμπορίου. Πολλοί από αυτού ανασυχούν για τι επιπτώσει στην απασχόληση ή τι επιπτώσει ε, τη πρόσβαση στα φάρμακα κανείς δεν αρνείται ότι να ανοίξει μια αγορά αυτό οδηγεί και σε βιομηχανική αναδιάρθρωση. Το πρώτο αποτέλεσμα είναι σαφώς ευεργετικό, αλλά κάποιοι χάνουν τις δουλειές τους, ενώ δημιουργούνται θέσεις εργασίας σε άλλους τομείς. Για το θέμα των φαρμάκων μπορέσαμε να τους ικανοποιήσουμε, για το σχέδιο συμφωνίας που συζητούμε συγκεκριμένα ορίζει ότι δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε καμία, κανένα περιορισμό της πρόσβασης ε, στα φάρμακα ή τα φαρμακευτικά προϊόντα. Στοιχείο που έχει ληφθεί σοβαρότατα υπόψη. Νομίζω, Πρόεδρε, ότι εν είδη συμπεράσματο πρέπει να πω ότι δεν θα πρέπει να φανταζόμαστε ότι η οικονομική ανάπτυξη οπουδήποτε μπορεί να λάβει χώρα χωρί δυσκολίε. Η δική μα οικονομική ανάπτυξη στη δική μα Ήπειρο δεν έγινε χωρί δυσκολίε. Όμω δεν πρέπει να υποτιμούμε και τι δυνατότητε τη ελεύθερη αγορά. Μπορεί να βγάλει του ανθρώπου από την φτώχεια. Όταν εργαζόμουν στο Χονγκ Κόγκ, στις ακτές της Κίνας τη δεκαετία του 90, είδα πως η άνοδος του ελεύθερου εμπορίου έβγαλε μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων από την φτώχεια. Φτώχεια στην οποία ήταν καταδικασμένη για δεκαετίες. Ο υπεύθυνο επίτροπο ε, είναι αυτή τη στιγμή στην Ινδία. Το έχουμε πει ότι θέλουμε μια συμφωνία μέχρι το τέλο τη χρονιά και θα πρέπει το σώμα μα να αποφασίσει ποια είναι η πορεία που θα ακολουθήσει. Πολύ ωραία. Ας ε, συζητήσουμε τώρα και με τα μέλη της δικής μας Επιτροπής. Να ξεκινήσω ρωτώντα εγώ, α, ρωτώντας κατά πόσον έχετε συμπεριλάβει τις γεωγραφικές ενδείξεις, τις προστατευόμενες γεωργικές ενδείξεις. Γιατί πριν από λίγα χρόνια όταν πήγα στην Ινδία μου έκανε εντύπωση το πόσο πολλά προϊόντα που πολλούνταν ήταν ε, φτιαγμένα στην Ινδία. Και εγώ ανακάλυψα ότι υπήρχαν ενοπνευματούχα ποτά, ενοπνευματώδη μάλλον ποτά της Ευρώπης, τα οποία κατασκευάζονταν όντως στην Ινδία. Ασχολείται λοιπόν με τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τις γεωγραφικές ενδείξεις η Επιτροπή κατά τη διάρκεια των ε, διαπραγματεύσεων. Ο Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν ήθελα να το πω, αλλά το θυμήθηκα όταν είπατε για αυτό το κρασί από την Ινδία. Πολύ ενδιαφέρον. Αυτό το ερυθρό της Ινδίας οδηγεί σε πολλές σκέψεις. Και είναι ενδιαφέρον να έχουμε αυτό το διπλό ρόλο μέσα σε αυτήν την επιτροπή αλλά και στην αντιπροσωπεία. Ε, η πρώτη φορά πήγα και άκουσα πώς ήταν η κατάσταση πριν και με εξέπληξε πάρα πολύ πόσο επέδρασε η συνήθεια της Λισαβόνα όσον αφορά το πώς μας υποδέχθηκαν οι Ινδοί εμάς στην αντιπροσωπεία. Ήταν πολύ διαφορετικά από την τελευταία φορά που πήγαμε. και Επομένω, αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα για τη συμπεριφορά, ακόμα και για τι ε, εμπορικέ διαπραγματεύσει. Και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε για την Ινδία ότι η Ινδία δεν είναι τελικά τόσο φτωχή. Είναι χώρα με πολλούς φτωχούς, αλλά ισχύει το αντίθετο γιατί μου δείξαν και κάποια μέρη που δεν ήταν καθόλου εκεί φτωχοί. Γιατί οι ομόλογοι μας είναι δεν ήθελαν να συζητήσουν, να συζητήσουν για θέματα εργασιακά, περιβαλλοντικά, κοινωνικής πρόνοιας. Όμως πολλοί συνάδελφοι σκεπτόμαστε ότι θα πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος. Αν όχι να συνδέσουμε τη συμφωνία με το περιβάλλον, τουλάχιστον να θέτουμε το θέμα όταν ε, εισάγουμε προϊόντα από την ιδέα τα οποία όμως έχουν παραχθεί με τρόπο που δεν θέλουμε, δηλαδή τα έχουν φτιάξει ανήλικοι. To forget those things, because if, if they are completely forgotten in that agreement, and I know it. Θα πρέπει να το επιθυμίσω αυτό στην Κομισιόν, μήπως τυχόν και το ξέχασαν. Γιατί ένα σωρό συνάδελφοι έχουν ασχοληθεί με αυτή την συμφωνία. Και άρα να μην το ξεχνάμε. Τέλειωσε σχεδόν, Πρόεδρε. Απλώς θέλω κάτι να αναφέρω όσον αφορά τους δασμούς. Να μην ξεχάσει η Κομισιόν. Να τώρα που στο πρώτο πρώτο που σας είπα. Να μην ξεχνά τους δασμούς για τα κρασιά. Πολύ σφιχτή αγορά στην Ινδία. Η δε παραγωγή Οι Ευρωπαίοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ να μπορούν να διεισδύσουν εκεί. Νομίζω θα, θα έχουν καλέ προοπτικέ. Ο κύριο Κάζακ, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή αυτό που μα είπε ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή για την φάση στην οποία έχουν φτάσει οι διαπραγματεύσει με την Ινδία. Επίση, με προσοχή άκουσα και τον κύριο Βότσον από την Αντιπροσωπή Ευρωπαϊκή Ένωση Ινδία παρά το Ευρωκοινοβούλιο. Νομίζω ότι υπήρξε μια ελαφρά απόσταση μεταξύ των όσων ακούσαμε και των όσων προσδοκούμε από μια τέτοια συμφωνία. Ο κύριος Βότσαν μας είπε ότι η δική πλευρά είναι πολύ αρνητική προς στιγμή στο να διαπραγματευτούν, πόσο μάλλον να συμπεριλάβουν πτυχές που ξεπερνούν το εμπόριο. Δηλαδή, περιβαλλοντικά, κοινωνικά ζητήματα, πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το καθεξής. Ο κύριος Μπερσέρο όμως μας είπε ότι αν η ειδική πλευρά μετακινηθεί θα πρέπει και εμείς να είμαστε σε θέση κάτι να παραχωρήσουμε. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει ένας, ε, ένας αέρας φιλοδοξίας ό,τι αφορά τις... αισιοδοξίας μάλλον ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις με την Ινδία. Και ο κύριος Δεχούφτ είπε μας εξέφρασε την θεώρησή του ότι ενδεχομένως οι διαπραγματεύσεις να έχουν ε, φτάσει σχεδόν στο τέλος τους ε, στη μέχρι τη συνοδοκορυφή Ινδίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ινδία. Αυτή η αισιοδοξία λοιπόν ε, για πού οφείλεται ήθελα να ρωτήσω. Μήπως έχετε κάποιες ενδείξεις από την πλευρά της Ινδίας μας ανησυχεί ιδίω αυτός προς από την πλευρά των ε, Ευρωβουλευτών και σε ό,τι αφορά κυρίως τα γενώσιμα φάρμακα. Το ανέφερε ο κ. Ντεχούχτ ότι υπάρχουν πολλοί φόβοι, πολλές ανησυχίες, όχι μόνο από την πλευρά των ειδικών συλλόγων, αλλά και από την ε, οργάνωση για τριχωρή σύνορα. Δεν θα πρέπει να ανησυχούμε ότι μπορεί να υπάρξει αρνητικό αντίκτυπο από τη συμφωνία αυτή στα γενώσιμα φάρμακα. Ευχαριστώ. Um, Θα είμαι και εγώ σύντομος. Μία παρατήρηση γενική, μακροπαρατήρηση αν μπορώ να την πω έτσι. Η Ινδία έχει κληρονομήσει από τη Βρετανία ένα πολύ καλό σιδηροδρομικό δίκτυο, το κράτος δικαίου και ούτω καθεξής. Όμως έχουν εισάγει και τον σοσιαλισμό και αυτό οδήγησε στο να δημιουργηθεί μια κλειστή οικονομία ο κύριος Βότσον που γνωρίζει τα πάντα εδώ, ίσως να μην γνωρίζει ότι τη δεκαετία του 60 υπήρχαν αυτά τα εκπληκτικά στατιστικά δεδομένα ότι οι εξαγωγές από τη Βρετανική και του Χονγκ Κόνγκ με πληθυσμό περίπου 4 εκατομμύρια ήταν πολύ υψηλότερες από τις εξαγωγές της Ινδίας με ένα πληθυσμό περίπου ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους. Αυτό γιατί οι Ινδοί φροντίζουν η οικονομία τους να είναι κλειστή, παράγουν προϊόντα τα οποία δεν είναι αντικείμενο εμπορία στην παγκόσμια αγορά. Δεν ήταν αυτό που ήθελα να πω. Όχι. Ο ο, ναι- ο Νεχρού και η οικογένειά του εισήγαγαν τον ε, σοσιαλισμό τη δεκαετία του 40. Ε, Αυτό ήθελα να καταστεί σαφές. Αυτή ήταν η γενικότερη μου παρατήρηση τώρα για θέματα ως πως τα περιβαλλοντικά πρότυπα, η παιδική εργασία. Ο τρόπος να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά είναι να υπάρξει μια, ελεύθερη, μια συμφωνία ελεύθερου, ελεύθερου με την Ινδία και πρόσβαση στην ε, αγορά τους. Τώρα, μια παρατήρηση γενική που ήθελα να κάνω και συνήθω κάνει ο εξαίρετο συνέδελφο ο κύριο Μάρτιν όταν ε, κάνουμε τέτοιε συζητήσει και θα το καταλάβει ο κύριο Γότσον. Ω Βρετανό βουλευτή έχω σοβαρέ ανησυχίε και εκφράζω νομίζω όλου του ε, ε, συναδέλφου από τη Βρετανία. Νομίζω ότι θα πληγεί ιδίω το σκοτσέζικο ουίσκι εδώ από μια, τη σύναψη μια τετοια συμφωνια Θα ήθελα λοιπόν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί επί του θέματος. Κύριος Νιούτον Ντάνε, Είμαι μέρος της αντιπροσωπείας κύριε Πρόεδρε, γι' αυτό και είμαι εδώ. Καταρχήν, Νομίζω ότι είναι πολύ προς ε, συμφέρον μας και συμφέρον της Ινδίας να ε, συναλλασσόμαστε. Είμαστε οι δύο μεγαλύτερες δημοκρατικές περιοχές ε, του κόσμου και θα ήταν τραγικό να μην συμφωνήσουμε. Όπως είπε ο Γκράχαμ και άλλοι από τους συναδέλφους, Μία από τις διαφορές θα είναι όταν θα φτάσουμε στο σημείο όπου αυτό το κοινοβούλιο θα χρειαστεί να κυρώσει μπορούμε να δεχθούμε ή να απορρίψουμε αυτή τη συμφωνία. Και πολύ σωστά οι συνάδελφοι είναι προσιλωμένοι στα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα θέματα που δεν είναι υποχρεωτικά εμπορικά. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι εάν δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα οι θα πρέπει να θέσουμε προϋποθέσεις αλλά οι δεν, δεν θα το δεχτούν και θα έχουμε πρόβλημα. Είναι ένα πολύ ε, υπερήφανο κράτος εκατοντάδων ετών και ε, θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε πάει ε, σε ένα χωριό στο Χιντεραμπάντ που ε, κατεργήθη η σκλαβιά των ε, παιδιών και μπορούσαν τα παιδιά να πάνε σχολείο αλλά υπάρχουν εκατοντάδες άλλων περιοχών όπου τα, υπάρχει εργασία παιδιών και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ε, φύρμωσε ο, ο Νεχρού. Εσύ είπε ότι ήταν του Νεχρού ενώ η εργασία των παιδιών υπάρχει ε, εδώ και ε, εκατοντάδες χρόνια στην Ινδία και δεν πρόκειται να αλλάξει ό,τι και να κάνουμε. Οπότε ε, σε μία συνεδρίαση ήμουνα δίπλα σε έναν ε, ε, δικηγόρο της αντιπολιτεύσεως και ο οποίος είπε κάτι πολύ έξυπνο ότι εσείς οι Ευρωπαίοι δεν χρειάζεστε τις ρήτρε αυτές απλούστατα επιμείνετε και πέστε ότι η Ινδία θα εφαρμόσει την δικιά της νομοθεσία διότι υπάρχει, απλούστατα δεν την υιοθετούν και αυτό θα επαρκέσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. δεν ε, μπορώ ε, να αντισταθώ ε, και να μην πω ότι όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας Ινδίας είναι πολύ ενεργά διότι είχαμε επισκεφθεί και τη χώρα πρόσφατα. Πρόκειται για μια κλειστή οικονομία η οποία ανοίγει γρήγορα και ε, βλέπουμε ε, ότι υπάρχουν θέματα τα οποία δεν αντιλαμβάνεται η Ευρώπη. Είναι μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται και εμείς απλώς μπορούμε να τους ζηλεύουμε αυτή την εποχή. Οπότε προς όφελος των πολιτών ε, της Ινδίας και της Ευρώπης θα είναι σκόπιμο να έχουμε ε, συμφωνίες ε, ελευθέρου εμπορίου που να είναι προς όφελος και των δύο περιοχών διότι θα δούμε ότι ε, εάν δεν υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις και όταν υπάρχουν απλώς εξαιρέσεις οι οποίες είναι αναπόφευκτες τότε θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο και τέλος θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε όλες τις πτυχές της συνδικής οικονομίας και της κοινωνίας χωρίς να ξεχνάμε ότι εδώ μιλάμε για μη, έναν πολιτισμό χιλιο, χιλιετηριών και η πρώτη μας προσπάθεια πρέπει να είναι να κατανοήσουμε καλύτερα και όχι υποχρεωτικά να, να καταδικάσουμε τους Ινδούς. Ευχαριστώ. Είναι 6 και 10, οπότε δεν δέχομαι ε, άλλα σχόλια και θα δώσω το λόγο στο Χέλμουτ Σότς απλώς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν μπορώ βέβαια να ανταγωνιστώ με τις παρατηρήσεις των Βρετανών αλλά μακροοικονομικά όταν κοιτάμε αυτή τη συμφωνία πρέπει να αντιληφθούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη πρόκληση και θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα οικολογικά θέματα και τα θέματα των ε, ανθρώπων ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά θα ήθελα να σας πω από πλευράς της Επιτροπής τα δύο θέματα τα οποία ήδη είχαμε, είχαν προκύψει σε σχέση με άλλες συμφωνίες. Όταν δηλαδή συζητούσαμε με την FTA και την ε, Κορέα είχαμε διαπιστώσει ότι στο άρθρο 35 του σχεδίου θα περιλαμβάνεται και πάλι μέτρα τα οποία δεν έχουν σχέση με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε μεταφέρει. Οπότε έχουμε θέσει αυτό το θέμα και υποθέτω ότι δεν είναι πολύ σοβαρό, δεν χρειάζεται δηλαδή να περιλάβουμε και πάλι αυτό το θέμα και εγώ θα ήθελα να είμαι σίγουρος ότι υπάρχει διαφάνεια. Έχουμε αναφερθεί στο θέμα των γενοσύμων φαρμάκων και πρέπει να πω ότι αν η Ινδία είναι ο πιο σημαντικός παραγωγός γενοσύμων φαρμάκων τότε θα δημιουργηθεί ένας φραγμός ε, στο εμπόριο και είναι κάτι το οποίο δεν είναι αποδεκτό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τρίτον θα ήθελα να πω ότι όταν ασχοληθήκαμε με τη Συμφωνία ε, ε, Ελευθέρου Εμπορίου ιδίως όσον αφορά την παραγωγική του γάλατος ότι το σενάριο θα οδηγήσει στην καταστροφή της γεωργίας αυτής. πράγμα το οποίο δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθεί η Ινδία και να είναι να είναι ε, αυτάρκης για θέματα που είναι πολύ βασικά για την χώρα αυτή. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα υπάρξει άλλη δυνατότητα και δίνω τον λόγο στην Επιτροπή για να μας παρουσιάσει ό,τι θέμα έχει. Ευχαριστώ κύριε Μορέρα, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και θα αναφερθώ στα συγκεκριμένα θέματα που ετέθηκαν. Είναι ένα από τα σημαντικά θέματα και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει η Ινδία να δεχθεί την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων ε, και ε, ακόμη και εκτός του γεωργικού τρομέα που είναι ένα βασικό θέμα. Ε, μία από τις πρώτες προτεραιότητες τις οποίες είδαμε και όπου θα υπάρξουν δυσκολίες ε, είναι η Γεωργία αλλά και εκεί παρακολουθούμε όσο καλύτερα μπορούμε. Ε, υπάρχει μία ε, μία επιστολή από τους γιατρούς χωρίς σύνορα προς τον κύριο Ντεγκούχτ όπου συζητείται το θέμα των, της πωλήσεως από την Ινδία των γενοσύμων φαρμάκων και εάν υπάρξουν και άλλα θέματα θα, τα οποία σας ενδιαφέρουν ευχαριστώ να σας απαντήσω. Βεβαίως ε, με κάθε τρόπο δεν πρέπει ε, να αντιταχθούμε στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και τέλος όσον αφορά τα δύο βασικά θέματα το περιβαλλοντολογικό και το κοινωνικό κάθε, σε, κάθε ευκαιρία εξηγήσαμε γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν θέλουμε να υπάρχει προστασία και ε, Πιστεύουμε ότι σαν όριμες δημοκρατίες η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ε, ε, και η δύο θα μπορέσουν να επιλύσουν τα προβλήματά τους σε ένα συμβιβαστικό πνεύμα και από τις δύο πλευρές και θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το θέμα αυτό. Και τέλος, όσον αφορά τον Οκτώβριο, ο Οκτώβριος ε, είναι βασικό ε, χρόνος για να μπορέσουμε να λύσουμε ορισμένα θέματα διότι διαφορετικά δεν βλέπουμε πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε από εκεί και πέρα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ε, θα έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα αλλά ελπίζουμε ότι μέχρι τότε θα μπορέσουν οι διαπραγματευτές να ολοκληρώσουν ολοκληρώσουν ορισμένες συζητήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι προς όφελος όλων και θα σταματήσω σε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ. Ας προχωρήσουμε στο σημείο 16 της ημερησίας διατάξεως μέσα εμπορικής άμυνας. Είναι ένα βασικό θέμα και θα ήθελα να σας πω ότι όποιος θέλει να φύγει να το πράξει όσο το δυνατόν πιο προσεκτικά κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε ε, ήσυχα και ήρεμα τη συζήτησή μας. Κύριε Ντάρτμουθ. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι θέματα ε, εμπορικής άμυνας, είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν και εντωμεταξύ έχουν προκύψει ορισμένες ε, περιπτώσεις που μας έχουν απασχολήσει στον τομέα αυτό μία πρώτη περίπτωση ε, αναφέρεται στην Κίνα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει την συζήτηση επί του θέματος και θα ήθελα να ξέρω εάν υπάρχουν ε, ε, εξελίξεις στο θέμα για να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε στην εποχή μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας Δίνω το λόγο στον υπεύθυνο για 8-10 λεπτά. για να μπορέσει να μας ε, κάνει μια εισαγωγή επί του θέματος. Ευχαριστώ κύριε Μορέρα. Αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε ορισμένα γενικά σχόλια, μετά θέσατε ορισμένα θέματα ε, και μετά ε, αναφερθήκατε στις μεταρρυθμίσεις. Καταρχήν, Πιστεύουμε ότι για να υπάρχουν κανόνες και να τους σεβόμαστε σε αυτή την περιοχή είναι κάτι πολύ σημαντικό για το σύστημα και οι πρόσφατες οικονομικές δυσκολίες είδαν ότι ε, η προσέγγιση δεν ε, μας καλύπτει είδαμε ότι υπήρχε φόβος πέρυσι ότι θα υπήρχε ένα τσουνάμι, ένα κύμα παλιριακών νέων περιπτώσεων και είναι ευτυχές ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη ε, αυξήθηκε, ε, φοβόμασταν μία αύξηση των περιπτώσεων την οποία όμως δεν διαπιστώσαμε και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε από τη βιομηχανία το γεγονός ότι ε, το σύστημα εμπορικής άμενας λειτουργεί σωστά έχει αποφύγει ε, τις, ε, τα προβλήματα άρα υπάρχει ένα σωστό σύστημα και τα μέσα τα οποία υπάρχουν μπορούν να εξεταστούν. Πάντως το μήνυμα το οποίο έχουμε εδώ είναι θετικό. Εσωτερικά έχουμε αναφερθεί στην ποιότητα του τι κάνουμε, πράγμα το οποίο ήταν πολύ σημαντικό και εσωτερικά έχουμε ε, καταρτήσει ένα σημαντικό πρόβλημα για να σταθεροποιήσουμε την ε, ποιότητα του τι κάνουμε και να διασφαλίσουμε ότι ε, τα θέματα θα αντιμετωπιστούν σαν παράδειγμα από όλους τους εμπορικούς εταίρους και ε, είδαμε ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να εφαρμοστεί η πολιτική αυτή ε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με αυτά τα εισαγωγικά σχόλια νομίζω ότι ξέρετε γενικώ τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής και ε, υπάρχουν και ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες ε, έχουν ε, επίσης εξεταστεί και αναφέρονται σε συστηματικά θέματα δηλαδή όπως διαπιστώσατε τώρα υπάρχουν ε, ορισμένοι ανταποδοτικοί δασμοί που νομίζω ότι έχουν εφαρμοστεί εις την ε, δημοκρατία της Κίνας και το ερώτημα είναι αυτό προκάλεσε κάποια αλλαγή υπάρχει αλλαγή αλλαγή πολιτικής. Όχι, διότι αν υπήρχαν τεκμηριωμένα θέματα και αν ε, η βιομηχανία μπορούσε να βρει ε, ότι ε, αποδείξεις ότι όντως υπάρχουν αυτές οι επιδοτήσεις θα ήμασταν πιο επιτυχημένοι αλλά η πρώτη αυτή περίπτωση δημιούργησε ορισμένα ερωτήματα με τους Κινέζους ομολόγους μας αλλά τώρα έχουμε συμφωνήσει ότι θα γίνει σωστά η έρευνα και θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα άπαξ και έχουμε συγκεκριμένα από τα γεγονότα. Έχουμε μία περίπτωση με τα υποδήματα και πρέπει να δούμε τι γίνεται στον τομέα αυτό. Για να σας υπενθυμίσω Είχαμε ε, επεκτείνει τα μέτρα αυτά για 15 μήνες διότι είδαμε ότι τα μέτρα αυτά όπως άλλωστε και τα αρχικά ε, δεν είχαν πολύ αποτέλεσμα αλλά χαιρόμαστε γιατί η Κίνα ακολουθεί τον σωστό μηχανισμό για την επίλυση των διαφορών στη Γενέβη. Εμείς είμαστε πολύ αισιόδοξοι για την περίπτωσή μας και θα δούμε τι, πού θα καταλήξουμε αλλά νομίζω ότι η περίπτωση αυτή έχει παρουσιαστεί πολύ σωστά και η ε, οι δικηγόροι μας ε, ε, διαβεβαιώνουν ότι θα κερδίσουμε. Υπάρχουν ε, συστηματικές επιτυχίες και νομίζω ότι όπως και στο παρελθόν και στο μέλλον θα είμαστε επιτυχείς σε αυτές τις περιπτώσεις. Όσον αφορά την ανάλυση της καταστάσεως σε σχέση με την Κίνα, θα συνεχίσουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ορισμένα κριτήρια και ε, θα προχωρήσουμε στα τεχνικά. Η συνεργασία με την Κίνα είναι καλή και τώρα εξετάζουμε τα λογιστικά. Ξέρετε ότι αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα. Πρέπει να μπορέσουμε να βασίσουμε τις αναλύσεις μας σε αξιόπιστο ε, στοιχεία και πρέπει να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή των λογιστικών κανόνων στην Κίνα για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε με τους Κινέζους ομολόγους μας και να δούμε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη και ιδίως σχετικά με την αξιολόγηση αυτή. Όσον αφορά την αναθεώρηση του PDI καθυστερεί. διότι υπάρχουν ενδιαφερόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διότι οι κανόνες στη Γενέβη δεν έχουν σταθεροποιηθεί και είμαστε ακόμη στην διαπραγμάτευση των κανόνων στη Γενέβη. Πρέπει ακόμη να καταρτήσουμε το πλαίσιο και ε, είμαστε υποχρεωμένοι να καθυστερήσουμε τη συζήτηση και γι' αυτό ακόμη βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Βεβαίως δεν έχουμε μείνει αμετακίνητοι η πολιτική είναι ένα σύνολο κανόνων και η εφαρμογή των κανόνων αυτό Και όπως είπα και προηγουμένως, με, σχετικά με την εσωτερική μας αξιολόγηση έχουμε εφαρμόσει τους κανόνες μας έχουμε δει ότι υπάρχουν και άλλες πολιτικές τις οποίες παρακολουθούμε Υπάρχει ένα πρόγραμμα αξιολόγησης της ποιότητας. Έχουμε ένα πρόγραμμα για τις παραγωγικές βιομηχανίες και ένα για τη βιομηχανία υπηρεσιών για να παρακολουθούμε όλα όσα γίνονται, ο, ο τρόπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε και θα σας παρουσιάσω συνέχεια μία πιο λεπτομερή παρουσίαση. Όσον αφορά το TDI, τις ε, επιπτώσεις της ε, συνθήκης της Λισαβόνας, ε, ξέρω ότι ο Επίτροπος ήρθε σε επαφή με σας καθηγητή Μορέιρα και ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα υπάρξει περισσότερη ευκρίνεια σε αυτό το τομέα. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ για όσο μας εξηγήσατε, για όσο μας ενημερώσατε όσον αφορά τα θέματα, τα σχετικά με